po' di ritardo dovuto... ελαφριά καθυστέρηση, μέχρι να μαζέψουμε τα μέλη της Επιτροπής, ε, ξεκινάμε με τις εργασίες. Ε, θα... Πρώτο σημείο είναι το σημείο 22 της Μεσής Διατάξεως. Θα ήθελα να σας προτείνω να εξετάσουμε ομού τις 22, 23, 24 και 25 αναφορές, διότι αφορούν στο ίδιο θέμα. Έχουμε και τον ίδιο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα απαντήσει σε αυτές. Ας ακούσουμε λοιπόν τους αναφέροντες και μετά τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια διαφωνία Πρόεδρε, περίμενα πως θα ανακοινώνατε στα μέλη της Επιτροπής ε, σχετικά με τις αποφάσεις ε, που λάβατε στο πλαίσιο των συντονιστών. Έχετε απόλυτο δίκιο, εντάξει. Θα επανορθώσω. Επειδή έχουμε καθυστερήσει, έλεγα μήπω ε, αυτές τι ανακοινώσεις τις έκανα στο τέλο, Το συγγνώμη από τους ε, αναφέροντε, ε, και θα πρέπει πρώτα να ενημερώσω την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της συνεδριάσεω των συντονιστών. Εξετάσαμε πρώτα απ' όλα το ζήτημα που αφορά στο ζήτημα της αναφοράς για τα αμόχωστο. Αυτό το θέμα το εξετάσαμε και στο Προεδρείο αλλά και στην Επιτροπή και αποφασίσαμε να την συμπεριλάβουμε στην μέση διάταξη τη προσεχού συνεδριάσεως της Επιτροπή μας με παράλληλη ακρόαση του Δημάρχου ε, Γαλανού και του αναφέροντος. Επειδή το ζήτημα είναι ιδιαίτερα λεπτό, το αποφασίσαμε η διεξαγωγή αυτής τη ακρόασης να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Επίσης ε, καταγράψαμε το θέμα των αποφάσεων που είχαμε λάβει στο παρελθόν ως Επιτροπή και για την ε, υποβολή δύο εγγράφων. Ένα έγγραφο αφορά τις κρατικές γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές για τις εργασίες της Επιτροπής και ο άλλος είναι ο κωδικός χρηστών πρακτικών. Αυτά και τα δύο έγγραφα έχουν διανεμηθεί. Αυτό μου το βεβαίωσαν όλες οι πολιτικές ομάδες που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οφείσαμε να αφήσουμε μια περίοδο προβληματισμού η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδριάσης της Επιτροπής μα. Ε, μετά από προτάσεις που θα υποβάλουν οι πολιτικές ομάδες για να καταλήξουν σε έναν κανονισμό πιο αποτελεσματικό που θα αφορά στις εργασίες ε, της Επιτροπής μας. Επίσης, ε, Αναφερθήκαμε στα δύο ζητήματα τα οποία έχουμε ήδη εξετάσει και εγκρίνει αναφορικά με τη διατύπωση γραπτών ερωτασιών τόσο για την ακρόαση των υποψηφίων στην θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσο για την ακρόαση των ε, νέων διορισμένων επιτρόπων των υποψηφίων. Ε, σκεφτήκαμε τρεις ερωτήσεις ε, στις οποίες ε, φυσικά θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν και κάποιες προτάσεις που θα υποβάλουν οι πολιτικές ομάδες. Ερωτήσεις συμπληρωματικές, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν, υποβληθούν τόσο στον υποψήφιο διαμεσολαβητή, όσο και στον υποψήφιο επίτροπο. Εγκρίθηκε λοιπόν αυτό το θέμα και οι ερωτήσει σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή. Η πρώτη είναι ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή στην προσεχή θητεία του, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία του γραφείου, τη υπηρεσία μάλλον του Δημοσιολαβητή και αν θεωρείται ότι χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού του καθεστώτου του Ombudsman και τι θα πρέπει να κάνουν οι αρχέ προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, των πολιτών. Και τρίτη, αυτές είναι τρεις ερωτήσεις. Λοιπόν, εμείς το σας τις διανύμουμε, τις ερωτήσεις αυτές, με ένα σημείωμα το οποίο θα κυκλοφορήσει μετά από το πέρας των εργασιών μας ε, τώρα. Σε ό,τι φορά την ακρόαση των υποψηφίων επιτρόπων, οι προτάσεις, οι ερωτήσεις μάλλον που πρότεινε η γραμματεία και που εγκρίναμε είναι τι συστάσει θέλει να κάνει ο αρμόδιος επίτροπο για τη βελτίωση τη διαδικασία η παραβάση που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη, πώς μπορεί η διαδικασία να ανταποκριθεί στις απαιτήσει των πολιτών και τρίτον ποιε είναι οι θέσει του Επιτρόπου σχετικά με μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών και μια διευκρίνηση σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα σε αναφορά και δικαίωμα ε, πρωτοβουλίες ε, με τη θέση σε ισχύ της Εθνικής της Αγώνας. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποστολή που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό στην Βουέλβα, αξιολογήσαμε τις δυσκολίες για υλοποίηση αυτής της αποστολής εντός του Δεκεμβρίου, διότι αφενός οι καθυστερήσεις με την οποία λάβαμε την άδεια σας υπενθυμίζω ότι το Προεδρείο χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να μας δώσει την εξοδότηση και ε, αφετέρου διότι έχουμε καθυστερήσει, καλέσαμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει περαιτέρω δράση και να μεταβεί επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο, χρήσιμο να σκεφτούμε πως η αποστολή μας στην Ουέλβα να διαξαχθεί μετά από αυτήν την ενημέρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί της εργασίας μας. Δυστυχώς ε, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε όλα τα σημεία τα οποία είχαμε σκεφτεί και είχαμε συμπεριλάβει στη μέσα διάταξη της συνεδριάσεως. Ε, η μοναδική πληροφόρηση που θα ήθελα να δώσω στα μέλη της Επιτροπής ε, είναι πως λάβαμε μια ανακοίνωση για την υλοποίηση διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων 2010 με, μέσα σε μια προθεσμία ιδιαίτερα σύντομη. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου να διατυπώσουμε προτάσεις ε, για δραστηριότητες ε, διακοινοβουλευτικές. Θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν, όπως κάλεσε και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ε, να υποβάλλετε αυτές τις προτάσεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρέωσεις μας. Ε, έτσι καθυστερήσαμε στην έναρξη των ε, εργασιών μας για 10 λεπτά και τώρα καθυστερούμε για περαιτέρω 10 λεπτά. Να σας συγχαρώ Πρόεδρε, διότι οι εργασίες σας ήταν ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικές ε, στο πλαίσιο της ομάδας των συντονιστών. και δεν είχατε φυσικά χρόνο να ολοκληρώσετε τις εργασίες. Αλλά έχουμε ένα σημείο στην μισή διάταξη, το οποίο υπήρξε μια πολύ σοβαρή παρατυπία, πολύ σοβαρή παρατυπία επαναλαμβάνω, την οποία θα ήθελα να ε, σας δηλώσω ότι εγώ ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου υπεύθυνο για τα θέματα πολυγλωσίας, δηλαδή μετάφρασης και διερμηνίας, θα ήθελα να θέσω το ζήτημα αυτό στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου και δεν θα ήθελα να το πράξω, διότι θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις, εάν προηγούμενα δεν το θίξω εδώ στην Επιτροπή σας και ιδιαίτερα σε εσά. Υπήρξε μία αναφορά, η οποία υποβλήθηκε από μία οργάνωση του Τολέδου, μια αναφορά όπως ε, τόσες ε, που φτάνουν στα χέρια μας. Εγώ θέλω να αξιολογήσω εδώ το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς. Ε, γεγονός είναι ότι αυτή η αναφορά εξετάστηκε από τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής μας και έγινε αξιολόγηση η οποία αναφέρει πως η αναφορά είναι απαράδεκτη και στα αυτή είναι μια αναφορά ε, που φυσικά έγινε στα ισπανικά και, και οι βουλευτές εν ώψη αυτής της αναφοράς ενεργούμε, ο κύριος Τουργκάης, εγώ και κάποιοι άλλοι, ενεργούμε λοιπόν ανακοινώνοντας την πόλη του Τολέδου, τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών ότι η αναφορά τους δεν έγινε δεκτή. Και με έκπληξη μετά από μερικές μέρες υπάρχει στα αγγλικά ανακοίνωση όπου αναφέρεται το, το αντίθετο. Λέγεται ότι ναι, έγινε δεκτή η αναφορά. Η αιτιολόγηση την οποία δεν γινόταν δεκτή, εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν ε, πολύ σωστή. Τώρα, και αυτό με οδηγεί σε δύο προβλήματα. Πρόεδρε. Πρώτον, κατά, ε, τόσο εγώ, ο κ. Τουρκάς και άλλοι συνάδελφοι, αλλά και άτομα της ε, ομάδας μου και της ομάδας του κυρίου ε, θεωρούμε ότι η παραδοχή ή όχι αυτής της ε, ε, αναφοράς θα πρέπει να εξεταστεί. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι παραδεκτή. Αλλά εν αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι να γίνονται σφάλματα διοικητικού χαρακτήρα και να εκδίδεται μία απόφαση ε, παραδοχής και μία ε, μη παραδοχής σε διαφορετικές γλώσσες. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη. Η γλώσσα στην οποία δηλώνεται η μη παραδοχή είναι αυτή που αφορά στους, τους ενδιαφέρομενους βουλευτές και αναφέροντες. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, βρήκαμε μία επιστολή δική σας την οποία φυσικά έγραψε η γραμματεία, ανακοινώνοντας στους αναφέροντες το αντίθετο από αυτό το οποίο οι βουλευτές είχαμε υποβάλει στις αρμόδιες αρχές της ε, πόλης του Τολέδου. Λοιπόν, σας ζητώ, όχι αυτή τη στιγμή, αλλά στην προσεχή μας συνάντηση, απαραίτητος να ε, θεωρήσουμε ότι να συζητήσουμε το θέμα και να μην να πούμε ότι δεν ε, κρίνουμε πως ε, πρέπει να γίνει παραδεκτή αυτή η αναφορά ε, εξ ονόματός της ομάδας μου, ο κ. Τουρκάζης από πλευρά του θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη και ότι η κρίση που αναφέρεται και και το αιτιολογικό της μη παραδοχής είναι πραγματικά άψογο και θέλω να σας ανακοινώσω ότι σε επίπεδο Προεδρείου του Κοινοβουλίου, εγώ ως Αντιπρόεδρος υπεύθυνο για αυτά τα ζητήματα της πολυγλωσσίας, θα θίξω το θέμα ώστε να εντοπίσουμε που, ε, υπάρχει το, που έγινε το λάθος και έτσι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα διότι αυτού του είδους τα σφάλματα δεν μπορούν, δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια διοίκηση σαν τη δική μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας και για την κατανόηση. Ευχαριστώ. Grazie, onorevole Ο κύριος Τουργκάης έχει το λόγο. Εν συντομία, Πρόεδρε, διότι το εξήγησε πολύ καλά ο συνάδελφος ε, Μιχαήλ Άγγελος Μαρτίνες, η κατάσταση είναι έκτακτη και εξαιρετική. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση έγινε αυτό το λάθος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και ως εκ τούτου πρόεδρε θα ήθελα να φυγεί το ζήτημα, δεν ξέρω, ίσως στην προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά απόψή μας είναι να μην δοθεί συνέχεια, να αρχιοθετηθεί λόγω αναφορά και να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε μάλλον, να μην ξανασυμβούν τέτοια λάθη, διότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ε, θίγουμε τις ε, εργασίες του Κοινοβουλίου μας. Ε, λοιπόν, σας ζητώ λοιπόν πρόεδρε εξ ονόματος της ομάδας μου, το έπραξε ο κύριος Μαρτίνης εξάλλου, εξ της του ομάδας, η αναφορά, η αναφορά, επαναλαμβάνω, να κλείσει και να αρχιοθετηθεί. Πρόεδρος. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα επί των οποίων δεν είχαμε χρόνο να, να συζητήσουμε κύριε Μαρτίνες. Πάντως το εγνώριζα το ζήτημα και άμεσα ζήτησα μια, έναν έλεγχο και απάντηση, μου δόθηκε μια απάντηση με κάποιο παράρτημα ε, ότι η υπηρεσία των μεταφραστών η μεταφραστική έλαβε, ανέλαβε την ευθύνη. Έχουμε ένα σημείωμα το οποίο μας εξηγείται το πώς συνέβη αυτό το θλιβερό γεγονός. Κάτι το οποίο πραγματικά στεναχωρεί όλους μας ε, και πρώτα απ' όλα εμένα. Το ζήτημα λοιπόν θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της ε, παραδοχής ή μη της ε, αναφοράς χρειάζεται δεχόμενα περαιτέρω αξιολόγηση γιατί εγώ δεν μπορώ έτσι αυτόνομα και καρδοδοκού να αποφασίσω ποια εκδοχή μπορεί να γίνει δεκτή, η ισπανική ή η αγγλική. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα να εξεταστεί ξανά στο πλαίσιο της Επιτροπής. Θα το ξαναθέσω στη συνεδρίαση των συντονιστών το ζήτημα για να απόφαση, αλλά η κατάσταση αυτή μας προσφέρει μια περαιτέρω ευκαιρία για να επαναλάβω προς ε, όλους ε, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει οργάνωση των εργασιών της Επιτροπής μας ε, τέτοια που θα μας επιτρέπει να αισθανόμαστε πιο κοντά στις εργασίες μας αλλά και να βοηθήσουμε και τους υπαλλήλους της Κομισιόν που έχει τεράστιο φόρτο εργασίες και μερικές φορές ενδέχεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Επ' αυτού λοιπόν έχει υπάρξει μια πρόταση αξιολόγηση της ε, παραγωγή ημί των αναφορών που θα μπορούσε να καταστήσει μετόχους όλους. Ξέρετε ότι περιοδικά ε, λαμβάνουμε αποφάσεις ε, περί των αναφορών. Εμείς εξετάζουμε μία προς μία στα έγγραφα που μας υποβάλλονται. Έχουμε ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν όμως αυτή την εργασία αρχίζουμε να την ε, αναθέτουμε σε εισηγητέ παραδείγματος χάρη, δηλαδή ε, κάποιους ε, βουλευτές μας, ε, ίσως έτσι θα μπορούσαμε να δίνουμε μια πρώτη απάντηση σε περιπτώσεις όπως αυτή που ακούσαμε και ελπίζω να μην επαναληφθούν ε, αν ε, λοιπόν έχουμε ικανοποιήσει το έτοιμά σας, ε, ξεκινάμε από το 22 με τα όσα είχα προτείνει, δηλαδή να εξεταστούν από κοινού οι αναφορές στα σημεία 22, 23, 24 και 25 που αφορούν και οι τέσσερις το θέμα της οδικής ασφάλειας στην Ιρλανδία. Και θα ήθελα να περάσω τώρα στην παρέμβαση του πρώτου αναφέροντα που αφορά στην, αναφορά 88-2009. Ο κύριος Σιον Φάρεν έχει το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να απευθύνουμε το λόγο σήμερα σε εσάς. Λέγομαι Σιον Φάρεν και είμαι εδώ με την σύζυγό μου και άλλες οικογένειες από την Ιρλανδία που χάσαμε τα παιδιά μας λόγω των προβλημάτων της οδικής σήμασης στην Ιρλανδία. Δεν μπορούν να διατηρήσουν μια ασφάλεια στους δρόμους οι αρχές αυτές. Για λόγους, γιατί η υποδομή ε, δεν είναι σωστή, δεν είναι σωστό το επίστρωμα που χρησιμοποιείται. Ε, έλλειψη ελέγχων ασφάλειας όταν για τη σιρήνηση των οδών η μη σύμβιβαση με τις κατευθύνσεις γραμμές και τα πρότυμα του Υπουργείου Μεταφορών, η έλλειψη υπολογιμότητας ε, για την ασφάλεια και η έλλειψη των, ε, της σωστής αντίδρασης της κυβέρνησης όταν υπάρχουν προβλήματα. Θα σας ε, παρουσιάσω τις κύριες περιπτώσεις της περίπτωσης ΣΥΝΑΤ που θα δείτε πώς τα σημεία 3, 4 και 5 χαρακτηρίζονται. Στις 12 Ιουνίου 2009 το αυτοκίνητο της έχασε τον έλεγχο περνώντας πάνω από μια καμπούρα του δρόμου που οφείλεται σε κάποιες εργασίες που είχαν κάνει οι αρχές εκεί. Υπήρχε μία μικρή, ε, μικρή μονάχα πινακίδα προειδοποίησης. Η Σινέατ ήταν μία πολύ ικανή ε, οδηγός. Πέρναγε Τρει-τέσσερι εβδομάδες από τον ίδιο δρόμο. Τον ήξερε λοιπόν καλά. Και ούτε η Κάρντε, ούτε το τοπικό συμβούλιο του Ντόνεγκαλ διατήρησαν την σκηνή του δυστυχήματος. Έβγαλαν απλώς σκουπίζοντας τα σκουπίδια που είχαν οδηγήσει στο δυστύχημα. Η Κάρτια επέστρεψε 23 ώρες μετά από το δυστύχημα, όταν είχε αλλάξει τελείως η σκηνή και εκεί πήρε φωτογραφίες και μέτρησε. Επίσης, δεν, δεν ε, δηλώθηκε ο θάνατος αυτός στον τόπο που είχαν εργαστεί. Εγώ δήλωσα το θάνατο της ΕΝΑΤ στην αρμόδια υπηρεσία τρεις μέρες μετά που έλαβε χώρα, χωρίς να γίνει καμία έρευνα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2006, πάνω από πέντε χρόνια μετά το δυστύχημα, μπορέσαμε να πείσουμε τις αρχές υγείας και ασφάλειας ότι έπρεπε να, ελέγξουν, να είχαν ελέγξει τις, ε, τους όρους προς τους οποίους έγινε αυτό το δυστύχημα. Γιατί θα έπρεπε να επιμένει η οικογένεια επί πέντε χρόνια για να τους πείσει για κάτι τέτοιο. Να τους πείσει δηλαδή ποια ήταν η, η υποχρέωσή τους, η ευθύνη τους. Το Συμβούλιο του Ανεγκαλ αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την νομιμότητα της έρευνας που έγινε από την Αρχή Ασφάλειας και Υγείας. Η έρευνα της Γκάρντια ήταν ελάχιστη. Μια ανεξάρτητη έρευνα έλεγε ότι θα πρέπει να γίνουν νέες έρευνες ε, και επερωτήσεις εάν χρειάζεται και ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2007. Και μόλις το Σεπτέμβριο 2009 μάθαμε ότι αυτή η ε, βρήκε ότι το Συμβούλιο του Νόνιγκαλ είχε κάνει σημαντικές παραλήψεις που οδηγούσαν σε μία παραβίαση του τμήματος 13 του σχετικού νόμου. Ορισμένα ανώτατα μέλη του Συμβουλίου του Τόνεγκαλ αποσύρθηκαν από την έρευνα. Ο διευθυντής όμως δεν, ο διευθυντής της ε, εισαγγελίας δεν ε, καταγγείλει και δεν ξέρουμε γιατί. Τα τελευταία 8 χρόνια είδαμε ότι πάρα πολλές υπηρεσίες, ε, το, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και πολλά άλλα δεν μας έδιναν πληροφορίες που ζητούσαμε συνεχώς και επιμόνως. Μέχρι σήμερα είδαμε κα πολλές ε, αρνήσεις, πολλές απορρίψεις, πολλές απαιτήσει ότι κανένας δεν έφταιγε, αλλά κανένας δεν μπορούσε να μας πει τι έφταιγε τελικά. Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ που διακυβεύονται για την κυβέρνηση της Ιρλανδίας, το λαό της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις καλύτερες μας προσπάθειες δεν μπορέσαμε να πείσουμε κανένα Υπουργείο να αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης. Κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει την κυβέρνηση της Ιρλανδίας να διορθώσει την κατάσταση και να υπάρχει ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο οι οικογένειες των ε, θυμάτων θα μπορούν να έχουν απαντήσεις στα προβλήματά τους. Προσπαθήσαμε να σας πούμε μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης, παραμένοντας ως των αντικειμενική. Πιστεύουμε ότι τώρα θα πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση. Προσπαθήσαμε να έχουμε απαντήσεις για τη δική μας περίπτωση, αλλά αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίγον και θα πρέπει να απαντηθεί. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο και να αποτρέψει κάτι τέτοιο να συμβεί στους άλλους. Εάν δοθούν ειλικρινείς απαντήσεις και υπάρχει το, η δυνατότητα να είναι κάποιος υπόλοιπος, θα μπορούμε εμείς να κλείσουμε την περίπτωση του θανάτου του Σινεάντου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μικάλα, αν θέλετε να δώσει κάποια άλλα παραδείγματα. λίγο με τον Μικάλη, είμαι... December 2004. Η κόρη μου σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2004. Θα ήθελα να σας πω ότι χρησιμοποιείται ένα ασφαλτόμιγμα, το DBM, στην οδοποιία των δρόμων της Ιρλανδίας ως μείγμα οδόστρωσης. Το μείγμα αυτό δεν δημιουργεί την απαραίτητη τριβή ανάμεσα στα ελαστικά των αυτοκινήτων και το δάπεδο. Φτιάχνεται από μία ελαφριά πέτρα η οποία διαβρώνεται εύκολα, λιένεται με την πάρδο του χρόνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την πάρδο του χρόνου η τελική επίστρωση χάνεται σιγά σιγά και αυτό οδηγεί σε πιο ολισθηρό οδόστρωμα. Το ζήτημα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε επιχείρημα σε προσφυγές που έχουν γίνει σε Ιρλανδικά δικαστήρια. Από ό,τι φαίνεται όμως οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το πυκνό αυτό ασφαλτόμιγμα, το DPM. Πριν από το 2006 έλαβαν ε, χώρα πάρα πολλά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τα οποία όμως ε, αποκρύφτηκαν, θα έλεγα, από τις ε, τοπικές αρχές. Στα πέντε χρόνια που πέρασαν μετά το θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα της Ashley, οι, οι αρμόδιες Ιρλανδικές αρχές για την οδική ασφάλεια δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία της οδικής ασφάλειας στην Ιρλανδία. Το όχημα, ο οδηγός, αλλά και το ίδιο το οδόστρωμα. Τα πρώτα δύο δεν ευθύνονταν για το θάνατο της Άσλεϊ. Το τρίτο όμως είναι ο βασικός λόγος που επήλθε το αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ο θάνατος της Άσλεϊ. Όσον αφορά τους οδηγούς, η Ιρλανδία έχει νέους πολύ αυστηρούς κανόνες για την πιστοποίηση των οδηγών, για τις άδειες οδήγησης. Επίσης είναι πάρα πολύ αυστηρή νόμοι όσον αφορά την οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ. Επίσης έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την αδειοδότηση οχημάτων. Όσον αφορά όμως την οδοποιία και το δόστρωμα, η, οδική, η αρμόδια Ιρλανδική Αρχή για την οδική ασφάλεια δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε τη και κανένα άλλο αρμόδιο φορέα στην Ιρλανδία δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του για την ποιότητα του, οδόστρωση. της οδόστρωσης. Οι τοπικές αρχές, οι οποίες θεωρούνται οι πλέον αρμόδιες, πολλές φορές παρακάμπτουν τους ελέγχους που κανονικά θα έπρεπε να γίνονται για τελικά που χρησιμοποιούνται στην οδόστρωση. Οι τοπικές αρχές μάλιστα δεν υπόκεινται καν σε ελέγχους. Το Δεκέμβριο του 2004 η κόρη μου η Άσλεϊ ενώ οδηγούσε οδήγησε πάνω σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που ήταν καλυμμένος με πυκνό ασφαλτόμιγμα DBM. Μάλιστα, η ε, οδική σήμανση, καθώς επίσης και η διαγράμμιση του δρόμου στο σημείο αυτό, δίναν την εντύπωση ότι ο δρόμος ήταν έτοιμος και ότι τα έργα είχαν ολοκληρωθεί, ενώ δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Προσπαθώντας να αποφύγει ένα αυτοκίνητο το οποίο έστρεβε προς τα δεξιά, φρέναρε, με αποτέλεσμα να έρθει σε σύγκρουση με ένα άλλο όχημα, το οποίο προσπάθησε να αποφύγει και εκτινάχθηκε όμως προς τα πίσω σε υπόσταση 30 μέτρων. Η Ashley δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και το όχημα το οποίο οδηγούσε είχε περάσει πρόσφατα από έλεγχο. Η οδόστρωση όμως πάνω στον δρόμο που οδηγούσε δεν ενδείκνυτο για καμία απολύτως ταχύτητα, ακόμα και για τις χαμηλές ταχύτητες. Η αρμόδια αρχή για την οδική ασφάλιση στην Ορλανδία έκανε έναν έλεγχο της κατάστασης και κατέληξε σε μία έκθεση. Η έκθεση όμως αυτή δεν μας ικανοποίησε χρειάστηκε να προσφύγουμε στο το δικαστήριο προκειμένου να καταλήξουμε σε μία απόφαση, προκειμένου να δούμε αν θα μπορούσε να κατηγορηθούν οι αρμόδιες Ιρλανδικές Αρχές Οδικής Ασφάλειας για το δυστύχημα αυτό. Το ότι δεν γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της οδοποίησης στην Ιρλανδία θεωρούμε ότι ήταν ο βασικός παράγοντας ο οποίος οδήγησε στο δυστύχημα αυτό. Είχαν ληφθεί αποφάσεις για την κατασκευή του δρόμου αυτού χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι και μάλιστα το δόστρωμα δεν είχε ολοκληρωθεί. Επίσης δεν είχε χρησιμοποιηθεί η επαρκής οδική σήμανση προκειμένου να φαίνεται ότι τα έργα δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί. Οι τοπικές αρχές δεν θεωρήθηκαν υπόλογες προς οποιονδήποτε υπουργό ή προς οποιανδήποτε κυβερνητική υπηρεσία για την κατάσταση στην περιοχή αυτή. Επομένως δεν φέρει κανείς την τελική ευθύνη. Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφύγουμε τέτοια άλλα δυστυχήματα στο μέλλον, προκειμένου να μην θρυνήσουν και άλλες οικογένειες. Μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια δυστυχήματα, αρκεί όμως να καταφέρουμε να α, φέρουμε τους υπόλοιπους στη δικαιοσύνη. Διαφορετικά θα έχουμε και στο μέλλον τέτοια δυστυχήματα, όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς μη ανάληψη ευθύνη στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει υπογράφησα τη δεύτερη ε, αναφοράς, η κυρία Κιν. Good morning. Καλημέρα σα. Λέγομαι Ρίτσαρ και Κέι Κιν. Ζουν στην ε, Κοντία του Καρή και στι 22 Απριλίου 2006 Ε, προσβλέπαμε στο μέλλον ε, μας ε, έχοντας έξι παιδιά, αλλά μέσα στις 24 ώρες, ώρες είδαμε ότι η κόρη μας Αελή σκοτώθηκε δραματικά σε ένα δυστύχημα οδικό στις 22 Απριλίου 2006. Ήταν επιβάτης σε ένα όχημα που οδηγούσε ο φίλος της 18 χρονών, γεμάτη ζωή, έτοιμη να αρχίσει σπουδέ τη, ε, να χαρεί τα ανήψια της, τις ανήψιές της. Το δυστύχημα έγινε σε ένα σταυροδρόμι, εκεί που λέγεται Ποροκρόρατοφ, στην κομιτεία του Κέρι. Εκείνη τη στιγμή των δυστυχημάτων αυτών ήταν αδύνατο βέβαια να καταλάβει κανένας το γιατί και πώς έγινε αυτό που έγινε. Γιατί η λύπη και η πίκρα είναι εκείνο που βαρύνει. Με το πέρασμα του χρόνου όμως μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε προσοχή μας στα τραγικά διαμεφόμενα της νύχτας αυτής και να δούμε ότι το δυστύχημα θα μπορούσε θαυμάσια να έχει αποφευχθεί προφανώς ποτέ δεν θα ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Γιατί τα δύο, οι δύο μάρτυρες ε, του δυστυχήματος σκοτώθηκαν ακαρέα και δεν υπέφεραν τουλάχιστον. Αυτό που είδαμε όμως ξεκάθαρα με την πάρα του χρόνου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία πιο ορθολογική προσέγγιση για την εφαρμογή των απαραίτητων ε, νόμων οδικής ασφάλειας σε όλο το δίκτυο των μεταφορών. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινοτική προσέγγιση για τη ζωστή έρευνα σημαντικών δυστυχημάτων στους δημόσιους δρόμους αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι νομοθετικές αρχές επανεξετάζουν τους ε, δικούς κανόνες και οδήγησαν αυτές οι προσπάθειες στη μείωση των δικημάτων, ιδίως των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Ε, χαιρόμαστε που τώρα πια δεν είναι αποδεκτή μια έτσι επιπόλαια προσέγγιση της ασφάλειας όσο ήταν στο παρελθόν δυνατόν να γίνει αυτό στην Ιρλανδία. Το γνώση μας τραγικής κατάστασης, ότι δεν υπήρχαν δηλαδή καθόλου καμία σήμαση, καμία πινακίδα στο σταυροδρόμιο αυτό και μπορούσε κανένας να περάσει χωρίς να γνωρίζει καν ότι υπήρχε ένα σταυροδρόμι. στο δυστύχημα της ε, κόρη μας ε, κρελήθηκε αμέσως η χωροφυλακή κάρτα, όπως και άλλες υπηρεσίες ε, του ανάγκης. Το σύστημα όμως που χρησιμοποιείται στην Ιρλανδία είναι όταν έρθει η Γκάρντια να δούνε κατά πόσον υπάρχει κάποιος εκεί που μπορεί να κατακορυθεί για το δυστύχημα, κάποιος αντίπαλος. Εάν όχι, δεν θέλω να πρέπει να κάνουν οτιδήποτε. Και τελικά η Γενική Συγγελία αποφάσισε ότι δεν θα υπάρχει κανένας κατηγορούμενος για το δυστύχημα αυτό. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Ε, η έρευνα που έγινε αφορούσε μόνο την καταγραφή του λόγου θανάτου. Τίποτα άλλο. Χωρίς να δίνει κανένα στοιχείο, χωρίς να μας βοηθά να κλείσουμε εμείς ε, την, ε, ε, το πένθος μας. Όσο μπαίναγε ο καιρό, προσπαθούσαμε να αναρωτηθούμε πώ έγινε το δυστύχημα και όσο πέρναγε ο καιρό, είδαμε ότι δεν ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν θύματα ε, τέτοιων δυστυχημάτων. Είδαμε ότι υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι βρισκόταν σε τόσο φοβερή κατάσταση πένθους για το ίδιο θέμα. Εμείς πάντα είχαμε κάποια ερωτηματικά για το ρόλο της τοπικής διοίκησης στην Κομιτεία του Κέρι. Κάποια στιγμή άρχισαμε να υποβάλλουμε ερωτήσεις και να συλλέγουμε πληροφορίες. Κατανοήσαμε την ύπαρξη της ε, Γκάρντα, ε, μια, ένα ε, έγγραφο 662, είναι ένα έγγραφο που συμπληρώνεται από την Γκάρντια μετά από δυστύχημα και ένα αντίγραφο θέλετε, στην Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας και στο τοπικό συμβούλιο της Κομιτείας του Κέρι. Εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το δούμε το έγγραφο αυτό, αλλά στην αρχή δεν μας το επέτρεψαν. Εμείς επεμέναμε, επιμείναμε και πήραμε ένα αντίγραφο και είδαμε ότι το αντίγραφο όμως, η έρευνα αυτή, η έκθεση αυτή, συγγνώμη, συμπεριλαμβάνει 11 σφάλματα. Το κυριότερο το κυριότερο σφάλμα ήταν ότι τοποθετούσαν το δυστύχημα αυτό 15 μίλια μακρύτερα από εκεί που έλαβε χώρα. Καταλαβαίνετε βέβαια πώς αισθανθήκαμε βλέποντας το έγγραφο αυτό. Ο φοβερός τρόπος με τον οποίο είχε καταγραφεί το δυστύχημα αυτό οδήγησε σε περισσότερες ερωτήσεις και συμπεράσματα ότι δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι υπήρχε προσπάθηση συγκάλυψης. Γιατί το σημείο που έγινε πραγματικά το δυστύχημα δεν είχε καμία σήμαση και καμία πινεκίδα. Δεν ξέρουμε σήμερα κατά πόσον αυτό συνέβαλε βέβαια στο δυστύχημα, γιατί δυστυχώ οι μόνοι που θα μπορούσαν να το πούνε ήταν ο οδηγό του οχήματο, ο οποίο επίση απέθανε, σκοτώθηκε. Μετά από 3,5 χρόνια εξακολουθούμε να ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρχές και τους νόμους που υπάρχουν. Δεν μπορούμε εμείς να προσφύγουμε κατά της Κομιτείας του Κέρι, ούτε φαίνεται ότι έχουμε το δικαίωμα να ενημερωθούμε λόγω περιορισμών μέσα στα πλαίσια δικής μας νομοθεσίας ελευθερίας ενημέρωσης σαν τελευταία προσπάθεια να εισακουστούμε, που βάλουμε την αναφορά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ο, πάρα πολλούς φακελούς πλήρης ε, ολυρογραφίας με όλα τα Υπουργεία, με όλες τις πληροφορίες που μας έδωσαν ή δεν μας έδωσαν. Έχουμε να εγγραφώ από την υπεύθυνη που λέει ότι πληρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομιτείας του Κερί και εκείνη αποφασίζει ποιος θα διωχθεί και ποιος όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την δραματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει κάποια, θα καταβάλει κάποια προσπάθεια για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή υποδομών στα κράτη-μέλη. Και το κεφάλαιο 7 της Οδηγίας 2006-082 για την ασφάλεια των οδών προβλέπει περιοδικό έλεγχο της ασφάλειας των οδών. Η υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας αυτής θα πρέπει να γίνει αμέσως και ε, να μην αναβληθεί η εφαρμογή της μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, όπως φαίνεται. Εμείς πιστεύουμε ότι κα... κάποια στιγμή θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του δικτύου ασφάλειας θα πρέπει να χθούν όλοι οι οδοί των κρατών μελών. Το κόστος των επιθεωρήσεων είναι μικρότερο από το κόστος των δυστυχημάτων σε πραγματικό και ανθρωπινό κόστος. Το πραγματικό κόστος μπορεί να υπολογιστεί. Το ανθρώπινο κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τα δίκτυα, τα οδικά αυτά να είναι κατά δυνατόν ασφαλή. Ο αξιολόγηση του κινδύνου και η πρόληψη είναι πολύ φτηνότερη από την αντιμετώπιση των δυστυχημάτων. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε μέτρο για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη ερευνούν σωστά δυστυχήματα που γίνονται στις δημόσιες οδικές ε, ε, οδούς. Αυτό που γίνεται στην Αδία είναι ανεπαρκές. Στην Ιρλανδία έχουμε ένα σύστημα όχι ε, νομικού, νομικής έρευνας, αλλά αντιπαράθεσης γιατί σε ένα δυστύχημα αναλαμβάνει την ευθύ η γκάρντα που έχει σαν στόχο να εξτάσει κατά πόσον υπήρχε μια εγκληματική πράξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικογένειά μας ήταν ακριβώς ότι κανένας δεν θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο και δεν θεωρεί κανένας ή οδήποτε υπεύθυνο. Δεν πιστεύουμε τη σωστή έρευνα όταν η οδηποτε υπευθυνο δεν πιστευουμε ότι σωστη έχει τον ηγετικό ρόλο. Αυτό μπορείτε να δείτε και με τον τρόπο που έχει συμπληρωθεί το CT66, το ερωματολογιό αυτό που προανέφερα. Γιατί, όπως σας είπα, το θέμα ε, που εξετάζει η Γκάρδια είναι κατά πόσον υπήρχε μια εγκληματική πράξη. Όταν ληφθεί αυτή η απόφαση, θεωρείται ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ευθύνη. Εμείς δεν κατηγορούμε την κάρτα συγκεκριμένα. Το σύστημα που έχουμε στο κράτος μας είναι εκείνο που είναι εσφαλμένο. Δεν είναι ένα σωστό ερευνητικό σύστημα. Αυτό που προτείνουμε είναι να ε, υπάρχει μία διαβουλευτική ερευνητική διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ε, εμπλεκόμενους σε ένα δυστύχημα, οικογένειες, μάρτυρες, εγκάρτια, όλες τις πτυχές ε, των δυστυχημάτων θα πρέπει να εξεταστούν με αυτόν τον τρόπο. Το σημερινό σύστημα είναι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις εκτός εάν έχει κάποιος εγκληματική νομική ευθύνη. Αυτό είναι απαράδεικτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συμβάλλει στην κατασκευή της υποδομής θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο να εξασφαλίσει η υποδομή που ε, προετοιμάζουν να εξυπηρετεί το στόχο τους. Ταυτόχρονα, οι τοπικές αρχές δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνε για τις έρευνες, γιατί πολλές φορές η μηχανική των τοπικών αρχών είναι εκείνοι που ελέγχουν το έργο τους. Οι ελλείψεις οδηγούν στην Ιρλανδία σε 10 θανάτους περίπου από δικά δυστυχήματα. Εμείς θέλουμε τώρα να υπάρχει δικαιοσύνη για την Αιλίν και τον Τρέβο και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να πετύχουμε. Δεν θέλουμε πληρωμές. Εμείς θέλουμε ευθύνες και συγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο μας έχουν συμπεριφτική μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε καμιά άλλη οικογένεια να μην περάσει από τον πόνο που ζούμε ακόμα και σήμερα. Θέλουμε μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο καθένας να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Εάν το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι καταγγελίες, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πραγματικά να γίνει. Αυτό σημαίνει να είναι υπόλογος κάποιος. Εμείς θρυνούμε το θάνατο της κόρης μας, Αιλίν, και του φίλου του Τρέβορ και δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά είδαμε κατόπιν ότι απλές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν απαντηθεί δεν απαντήθηκαν. Λόγω του συστήματος που υπάρχει στην Ελλαδία Πιστεύω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι πεθούσες οικογένειες να είναι εκείνες που θα μετράνε πιο πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ευρωπής. Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλω να μιλήσω για τις ε, αναφορές αυτές που έχουν να κάνουν με πολύ θλιβερά γεγονότα για τις οικογένειες αυτές, φοβερά επώδυνα γεγονότα. Ως ε, γονιός καταλαβαίνω τον θρήνο σας, καταλαβαίνω την απόγνωσή σας, την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τις αναφορές αυτές και να σας καθησυχάσω λίγο σε σχέση με αυτά τα οποία στοχεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Οι αναφορές αναφέρονται σε μία οδηγία του 2006, την 812 του 2006, όσον αφορά τη διαχείριση ασφάλειας των δικών υποδομών η οδηγία αυτή είναι μια πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά που υιοθετήθηκε το 2008 στις 19 Νοεμβρίου 2008 και όπως είπε και ένας από τους υπογράφοντες θα αρχίσει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2010 μόνο. Επομένως, ε, όταν επέλθει το αυτοκινηστικό δυστύχημα δεν ίσχυε η οδηγία αυτή, ήταν απλώς μια πρόταση την εποχή εκείνη. Ακόμα και αν ίσχυε βέβαια, δεν θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο γιατί ισχύει μόνο για τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα και όχι για τα εθνικά οδικά δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχει ο περιορισμός αυτός, λυπάται για τον περιορισμό αυτό, αλλά η οδηγία αυτή έχει να κάνει μόνο με τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα που αποτελούν βέβαια ένα μικρό τμήμα των οδικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θελήσαμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή οδηγία αυτή και σε άλλα τμήματα του οδικού συστήματος, των δικών υποδομών, αλλά δεν πετύχαμε κάτι τέτοιο. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι η εν λόγω οδηγία, μολονότι δεν έχει αρχίσει ακόμα να ισχύει, θα επιφέρει, πιστεύω, μια, θα δώσει μια απάντηση για τις τραγωδίες αυτές. Δηλαδή, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διεξάγουν έλεγχο δικής ασφάλειας και οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στα δυστυχήματα, στα ατυχήματα που έλαβαν χώρα. Επομένως, ε, κάποια διδάγματα τουλάχιστον θα αποκομιστούν από τις τραγωδίες αυτές, επαναλαμβάνοντας βέβαια πάλι ότι η οδηγία έχει να κάνει μόνο με τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα. Η 881 αναφέρεται στην ε, παραβίαση των κανόνων όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία. Εξετάσαμε την αναφορά αυτή, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε εδώ πέρα για ποιο λόγο γίνεται η αναφορά αυτή, εφόσον η οδηγία, όπως σας είπα, που αναφέρεται στην ε, αναφορά αυτή, έχει να κάνει με την προστασία των εργαζομένων και όχι με την ε, προστασία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της κοινοτική νομοθεσίας δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια ικανοποιητική απάντηση στις τραγωδίες αυτές που μας περιέγραψαν οι οικογένειες εδώ. Ολοκληρώνοντας πάντως θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα λίγο πιο θετικά Όσον αφορά τι μελλοντικέ πράξει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφώ ε, εμπλέκεται σαφώ πάρα πολύ στο θέμα τη διαχείριση οδική ασφάλεια και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιφέρει εδώ τη θέμενη αξία. Του χρόνου, το 2010, θα ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να κινητοποιήσει γύρω από το πρόγραμμα αυτό τα κράτη-μέλη με έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, δηλαδή να σώσουμε 20.000 ζωές στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα το στόχο αυτό, σχεδόν τον έχουμε πετύχει και βέβαια δεν τον πετύχαμε εξαιτία της διεύρυνσης περισσότερο, γιατί προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη όπου το επίπεδο της οδικής ασφάλειας ήταν πολύ χαμηλό. Έγινε όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμάζει αυτή τη στιγμή το τέταρτο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα καλύψει την περίοδο 2011 με 2020. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της διαβούλευσης για το πρόγραμμα αυτό και γίνεται διαβούλευση και με τους πολίτες, ξεκίνησε μέσω του διαδικτύου αυτή, και είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του 2009 και βέβαια κάθε πολίτης μπορεί να πάρει μέρος στη διαβούλευση αυτή, να εκφράσει την άποψή του. Οργανώνουμε και θα οργανώσουμε και άλλες συνεδριάσεις με όλα τα συμβαλώμενα μέρη για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε το νέο αυτό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καθοριστεί τα ακριβή στοιχεία του προγράμματος αυτού, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα βάση της διαβούλευσης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά έχει τεθεί ήδη μια σημαντική προτεραιότητα. Η προστασία των πιο ευπαθών ομάδων και πιο συγκεκριμένα η προστασία των νέων οδηγών Επιμένουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό και αποτελεί κέντρο, βασική προτεραιότητα του τέταρτου προγράμματο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχει εντοπιστεί ω βασικό πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία του προγράμματο αυτού θα μα δοθεί και η δυνατότητα να εξετάσουμε και κάποια από τα ερωτήματα και τι παρατηρήσει που τίθενται μέσω των αναφορών που ακούσαμε όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τις έρευνε που γίνονται μετά από κάποιο ατύχημα και όσον αφορά την, τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που θα πρέπει να γίνονται για τις οδικές υποδομές. Κυρία Πρόεδρε, μολονότι γνωρίζω ότι δεν δώσαμε συγκεκριμένα συγκεκριμένες απαντήσεις μέσω της φυστάμενης νομοθεσίας, αν μη τι άλλο, Πιστεύω ότι σας ε, καθησυχάσαμε κάπως για την μελλοντική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την οδική ασφάλεια και για την αποφασιστικότητα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούμε το ζήτημα αυτό και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας, αλλά ευαίσθητος δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα, σοβαρά προβλήματα τα οποία ακούσαμε Ακούσαμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους ε, που έκαναν κάποιες προτάσεις ε, προκειμένου να αποφευχθούν ε, περαιτέρω τραγωδίες. Πέραν της δικής τους τραγωδίας λοιπόν φροντίζουν να αποφευχθούν τραγωδίες στο μέλλον. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εσά και τα μέλη τη Επιτροπή Αναφορών που υποδέχτηκαν εδώ πέρα τι τρει οικογένειε και που τι άκουσαν τόσο προσεκτικά, καθώ περιέγραφαν τις, τα τραγικά αυτά δυστυχήματα των συγγενών τους, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαι όμως απόλυτα ικανοποιημένο με την απάντησή της. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις υφιστάμενες οδηγίες που έχουν μεταφερθεί σε εθνικές νομοθεσίες και οι οποίες απαιτούν ότι όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια ανεξαρτήτων των, ανεξαρτήτως των ε, έργων που γίνονται, των έργων οδοποίησης. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μα είναι ότι τρεις νέες γυναίκες που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται, να ζουν και να έχουν ακόμα και παιδιά, δεν ζουν πλέον. Έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην περίπτωση της ε, Αιλίν, όπως είπε και η μητέρα της και αδελφή της, στην περίπτωση της Αιλίν Κιν, βρέθηκε σε μία διασταύρωση, δεν υπήρχε καμία σήμανση και έπεσε αυτή την παγίδα του θανάτου και στην περίπτωση της άλλης οικογένειας, της ε, Ashley Gallagher, είναι μια κοπέλα η οποία πήρε το πτυχίο της, θα ε, πήγαινε προς μια τράπεζα για να πάρει ένα δάνειο για να πάει στις Ηνωμένε Πολιτείε. Άρχιζε πήρε το αυτοκίνητό της για να πάει προς, τη θάλασσα, ε, προς την ε, ε, τράπεζα αυτή, οδήγησε σε ένα τμήμα του δρόμου που ήταν καλυμμένο με το ασφαλτόμιγμα DBM, δεν υπήρξε καμία σήμανση για το όριο ταχύτητας και έχασε τη ζωή της. Οι τοπικές αρχές θεωρώ ότι είναι υπεύθυνε και θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο θάνατος των τριών αυτών κοριτσιών δεν οφείλεται στις κοπέλες αυτές, δεν οφείλεται στην οδήγησή τους δηλαδή, αλλά είναι ευθύνη των ε, τοπικών αρχών. Καμία ευθύνη δεν θα πρέπει να επιρριφθεί στις τρεις αυτές κοπέλες. Και μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, η πληγή αυτή θα παραμένει ανοιχτή και δεν θα καταφέρει να λάβει τέλος, αν θέλετε, το δράμα των τριών αυτών οικογενειών. Η ε, Επιτροπή των Αφορών θα μπορούσε να υποβάλει περισσότερο το ζήτημα αυτό προς την Επιτροπή των ε, Μεταφορών, της οποίας είμαι και εγώ μέλος. Και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε περισσότερο ποιες είναι οι επιδόσεις κάθε κράτους μέλους. Γιατί αν θέλετε, το πίνακα αξιολόγηση αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αυτό λοιπόν το οποίο σα ζητώ να κάνουμε ω Επιτροπή Αναφορών, να υποβιβάσουμε του φακέλου αυτού, τι αναφορέ αυτέ, στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τι τρει οικογένειε που ήρθαν στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα, καθώ επίση ε, και του Ευρωβουλευτέ που ασχολούνται με τι αναφορέ αυτέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή τη. Σίγουρα το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να λάβει υπόψη τη την δύσκολη ευαίσθητη αυτή κατάσταση. Μιλάμε εδώ πέρα για ανθρώπινες ζωές, αλλά μιλάμε και για νομικέ ευθύνες. Και νομίζω ότι η προσέγγιση ήταν θετική. Από ό,τι φαίνεται, η νομοθεσία στην οποία βασίζονται οι αναφέροντες θα αρχίσει να ισχύει τελικά το 2010 και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινωτική αυτή νομοθεσία θα αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα. Όπω είπα όμω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει δυνατότητα επέκταση του πεδίου εφαρμογή κοινοτική αυτή νομοθεσία, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι επιθεωρήσει τη ε, οδική ασφάλεια και προκειμένου τελικά να τροποποιηθεί η κατάσταση στο μέλλον και να δούμε μια ουσιαστική βελτίωση. ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια ουσιαστική απάντηση σήμερα στι οικογένειε που είναι εδώ μαζί μα, θα ξέρουν ότι κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν και αυτέ στο να καταλήξουμε σε μια κοινοτική νομοθεσία που θα συμπεριλαμβάνει και του ελέγχου αυτού. Και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθο, γίνεται και αυτή η διαδικασία διαβούλευση. Είναι μια διαβούλευση που αφορά και του πολίτε. Είναι μια ανοιχτή διαβούλευση που θα επιτρέψει και σε οικογένειε που είναι παρούσε σήμερα, αλλά και σε άλλου πολίτε να συμμετέχουν ενεργά και να υποβάλουν τι δικέ του ιδέε και τι δικέ του απόψει για το πώ θα πρέπει να διαμορφωθεί στο μέλλον το τέταρτο πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια. Σίγουρα δεν επιλύουμε το πρόβλημα εδώ σήμερα, αλλά αν μη τι άλλο επιτρέπουμε στου παρόντε να αισθανθούν ότι κατά κάποιο τρόπο συμβάλλουν και αυτοί. Υπόθηκε ότι από τον Τζίμ ότι θα μπορούσαμε να υποβάλουμε το ζήτημα και στην Επιτροπή Μεταφορών προκειμένου να ασκήσουν περισσότερη πίεση. Ίσως αυτό να ήταν χρήσιμο όντω. Και νομίζω ότι ενδεχομένω όντω θα μπορούσε να επιφέρει περισσότερη πίεση, γιατί αυτό που ζητούν και οι οικογένειε το είπαν ξεκάθαρα, είναι ότι θέλουν να αναγνωρίσουν οι τοπικέ αρχέ ότι είναι αυτές υπεύθυνε και ότι η ευθύνη δεν επιβαρύνει την Σινέν, την και την Άσλι, τις τρεις όμορφες αυτές κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους. Ακόμα και αν δεν μπορούμε εμεί επίσημα να πιέσουμε τις τοπικέ αρχές να, να λάβουν την ευθύνη αυτή ω Επιτροπή Μεταφορών και με την ε, υποβολή του φακέλου αυτού και στην Επιτροπή Μεταφορών θα καταφέρουμε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Η ε, κυρία Γκρουνή. ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συλληπιθώ τις οικογένειες, να τις ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Καταλαβαίνω πόσο επώδυνη είναι η όλη διαδικασία και εγώ με μητέρα καταλαβαίνω απόλυτα τον πόνο τους και κάθε φορά και εγώ τηλεφωνώ στις τρεις κόρες μου κάθε φορά δύο που παίρνουν το αυτοκίνητο προκειμένου να είμαι σίγουρο ότι έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι. Όταν ήμουν βουλευτή στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση ασχολήθηκα πολύ με τα ζητήματα αυτά της οδικής ασφάλειας που είναι πολύ σημαντικά, πολύ ουσιαστικά. Μιλάμε σήμερα για την κατάσταση των ε, δρόμων, μιλήσαμε επίσης και για την κατάσταση ιδιαίτερα των νέων οδηγών, ιδίως των οδηγών υπό την επίρρεια του αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Είναι πολύ σημαντικό ως ευρωβουλευτές να ασχοληθούμε με τα διαφορετικά αυτά ζητήματα. Και ακόμα και αν και σήμερα Βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχει μια ανεπάρκεια στις απαντήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς οικογένειες αυτές, ότι δεν μπορούν να δοθούν ουσιαστικέ απαντήσεις. Ας έχουμε κατά νου ότι οφείλουμε για όλες αυτές τις περιπτώσεις να δώσουμε λύσεις. Ας ασκήσουμε την κατάλληλη πίεση προκειμένου να κινηθούν τα πράγματα. Και ας έχουμε κατά νου ότι ε, η οδική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο και ότι πρέπει εμείς οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές να δείξουμε ιδιαίτερο θάρρος και σθένος κάθε φορά που ασχολούμε με αυτά. Μιλάμε πάρα πολλές φορές για το ζήτημα της ταχύτητας, του ορίου ταχύτητας, μιλάμε πάρα πολλές φορές για την κατάσταση των δρόμων. Η κατάσταση όμως των δρόμων συνδέεται πάρα πολύ με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επισέρχονται τέτοιοι παράγοντες. Δεν ταξιδεύω ίδια πάρα πολύ. Η κόρη μου όμως ήταν ε, φύγιο πέρα στην Λιμρίκ της Ιρλανδίας είχε πάει δηλαδή εκεί πέρα κατά τη διάρκεια μια συγκεκριμένη περίοδου για να ασχοληθεί με ένα παιδάκι και όντας εκεί για να την επισκεφθώ, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κατάσταση των δρόμων, το πόσο στενή είναι πάρα πολλές φορές οι δρόμοι, η ταχύτητα με την οποία τρέχουν πολλές φορές οι οδηγοί, το ότι πολλές φορές σε ένα πολύ στενό δρόμο, ενώ οδηγεί κανείς, φτάνουν πάρα πολύ γρήγορα από το αντίθετο ρεύμα λεωφορεία, Δεν λέω ότι στη Γαλλία είμαστε καταπληκτικοί, αλλά τουλάχιστον έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες. Δεν γνωρίζω βέβαια το σύνολο του δικού συστήματος στην Ιρλανδία, πάντως από τη σύντομη με αυτή η επίσκεψη κατάλαβα ότι σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο δικό εκεί σύστημα. Και αν καταφέρουμε εμείς να επιφέρουμε μια λύση υποβάλλοντας την υπόθεση αυτή, τις υποθέσεις αυτές στην Επιτροπή Μεταφορών, τότε συμφωνώ και εγώ να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας παρακαλέσω να είστε πιο σύντομοι. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, παρεμβάσεις ε, και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος κλπ. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλήξουμε κάποια συμπεράσματα το ταχύτερο δυνατόν για να ακούσουμε ενδεχόμενα και την απάντηση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τις οικογένειες που ήρθαν εδώ και να ευχαριστήσω και τον Κομισιόν που μας έδωσε μια ειλικρινή τίμια απάντηση. Και ελπίζω πραγματικά, όπω είπε η Κομισιόν, να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε. Αυτό που ανέφερε η οικογένεια Κίν ότι σύμφωνα με την νομοθεσία στην ε, Ιρλανδία, η Γκάρντα, η χωροφυλακή επιτόπου, εξετάζει ένα δυστύχημα μόνο υπό τη σκοπιά κατά πόσον έφταιγε κάποιος επιτόπου εγκληματικά, αν υπήρχε δηλαδή κάποια παράβαση. Εγκληματική. Αυτό είναι το κύριο θέμα, το οποίο πρέπει να αλλάξει. Κατά πόσο θα αλλάξει στην Ευρώπη ή στην Ιρλανδία δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξει πάντως. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ε, σημείο είναι ότι οι σήμανση των δρόμων είναι ε, ανεπαρκής. Ακόμη και στο δρόμο στον οποίο σκοτώθηκε η Άριν Κιν, έχουμε εδώ μια φωτογραφία ενός σήματος, μιας πινακίδας που έχει μπει χωρίς νόημα. Γιατί εδώ από τη φωτογραφία ξεκάθαρα φαίνεται ότι είναι σταυροδρόμοι. Ε, η πανηγίδα αυτή που εγκαταστήθηκε μετά το δυστύχημα δίνει την εντύπωση ότι είναι μια διασταύρωση σχήματος staff. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σωστή σήμαση, ακόμα και μετά από όλα αυτό που έγινε. Και θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Higgins, αν μπορεί να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών, οπότε θα προωθηθεί το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Onorevole Joy Higgins. Thank you, uh, Chairperson. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι συγκινούνται από τις μαρτυρίες που ακούσαμε σήμερα από τις οικογένειες Φάρεν, αλλά και εκείν Το να χάσει κανένας αγαπημένο του πρόσωπο από φυσική καταστροφή είναι πάντα δύσκολο. Το να γίνει κάτι τέτοιο από ένα τραγικό δυστύχημα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εάν όμως το δυστύχημα αυτό οφείλεται σε ένα αμέλεια των τοπικών ή κρατικών αρχών, είναι αβάσταχτο. Και πραγματικά θα ήθελα να εγκομιάσω τις οικογένειες αυτές που επέμειναν μετά από τους τραγικούς θανάτους των αγαπητών τους προσώπων τριών νέων γυναικών και ενός νέου άντρα. Νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογικό να αποζηθεί κανένα στη γωνιά του και να θρυμνήσει και χρειάζεται πάρα πολύ τόλμη για να εγκαταλείψει τη γωνιά αυτή. Σαν ε, μαρτυρία για εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και ιδίως να δείξουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη των αρχών και να προσπαθήσουν να ληφθούν δράσεις από τις τοπικές και εθνικές αρχές για να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον. Στην Ιρλανδία, στην ε, Ήπεθρο, έχουμε πολλούς στενούς δρόμους που δεν θέλουν να μετατραπούν σε αυτοκινητόδρομους. Από την άλλη μεριά όμως θέλουμε αυτοί οι δρόμοι να είναι ασφαλείς με τα σωστά οδοστρώματα από τις τοπικές αρχές, όπως ελέγχθη σήμερα. Είναι απαραίτητο αναγκαίο κάτι τέτοιο. Να υπάρχει σωστή σήμανση επίσης, ούτως ώστε οι τοπικές αρχές να κάνουν τα πάντα ούτως ώστε οι οδηγοί των οχημάτων να βρίσκονται σε μια ασφαλή κατάσταση. Και εάν υπάρχει τελικά δυστύχημα, τότε αυτό να οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα του οδηγού και όχι σε έλλειψη δράσης των αρχών. Και συμφωνώ με τους αναφέροντες όταν αναφέρονται στο θέμα του, της ευθύνης του να είναι κάποιος υπόλογος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν απαραίτητο κάποιον να καταδικαστεί, αλλά θέλουν να υπάρχει ευθύνη, ούτως ώστε να μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα και συμφωνώ με τον Τζιμ Higgins ότι ε, μια περαιτέρω έρευνα και δράση να ζητηθεί η συμμετοχή της Επιτροπής Μεταφορών. Από την άλλη μεριά, πραγματικά, οι εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι και οι εθνικοί βουλευτές στην Ελλοδία και σε κάθε κράτος μέλος έχουν μια πραγματική ευθύνη να εξασφαλίσουν να είναι επιτόπου συνεχώς, να εξασφαλίσουν οι υπάλληλοι των τοπικών αρχών τους να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και σαν αποτέλεσμα των μαρτυριών που ακούσαμε σήμερα, θα πρέπει να γίνει περισσότερο κατανοητό μεταξύ των εκλεγμένων εκπροσώπων ότι πρέπει πάλι των διαφόρων συμβουλίων να φροντίζουν να γίνεται ό,τι πρέπει, να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να αποφευχθούν αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίε στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κυρία Βαρτμάν. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την, ε, τα συλληπιτήριά μου και την ευαθιά μου στι οικογένειες αυτές. Θέλω να τις πω ότι θαυμάζω που τόλμησαν να έρθουν εδώ να μας παρουσιάσουν την υπόθεσή τους. Επί της ουσίας μπορώ να συμφωνήσω με τον προαλήσαντα. Θα ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο. Έχουμε όλοι δικαίωμα ενημέρωση και απορώ γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάπου ένα μέτρο, μία διάταξη που να προβλέπει ότι θα πρέπει στις οικογένειες των θυμάτων να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν που έδρασε ήδη, μήπως είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια μέθοδος ώστε να μην χρειαστεί να αγωνιστούν τόσο οι οικογένειες για να πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν. Ε, Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν νομίζω ότι θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα. Η επιθυμεί να Εντάξει, δεν χρειάζεται. Να ευχαριστήσω εκ νέου τους αναφέροντες ε, τις οικογένειες των θυμάτων που έφεραν ενώπιον μας ε, τις υποθέσεις αυτές. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να μεταφραστούν σε κάτι το πιο απτό. Εξετίμησα την ε, της πατρίς του κυρίου Higgins ε, που έκανε έκκληση στους αρμοδίους, στους υπεύθυνους ε, στην Ιρλανδία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αναλυθούν πρωτοβουλίες για να δοθούν απαντήσεις δυστυχώς σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. <clears throat> Φυσικά ένα αίτημα από όλες τις πλευρές, δηλαδή να προωθηθεί περαιτέρω αυτή η αναφορά προς την Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου Ζητήσουμε λοιπόν από την Επιτροπή Μεταφορών να εξετάσει το θέμα της οδικής ασφάλειας, ε, διότι η Ιρλανδία μέσω των μαρτυριών που ακούσαμε σήμερα κατέδειξε ότι έχει πάρα πολλές ελλείψεις, ε, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Ε, στη δική μου πρώτα απ' όλα στην Ιταλία υπάρχουν πολλές ελλείψεις και ζούμε παρόμοιες τραγωδίες. Δυστυχώς οι τοπικές και οι εθνικές αρχές δεν αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν το ζήτημα με καταλληλότερο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή να στείλουμε έτοιμα στις ε, Ιρλανδικές Αρχές προκειμένου να τους καταδείξουμε πως ε, το ζήτημα μας απασχολεί, μας ενδιαφέρει, να ζητήσουμε επαλήθευση της κατάστασης και να λάβουμε και απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που ετέθησαν ε, τώρα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω το εξή ε, κατανοώ την απάντηση που μας δώσατε και συμμερίζομαι με την ε, αναφορά ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κομισιόν, δεν αποτελεί αντικείμενο των οδηγιών που αναφέρθηκαν διότι είναι στήματα που αφορούν ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτών των οδηγιών. Λοιπόν όμως αυτές οι οδηγίες ε, ορίζουν κάποιους κανόνες ε, αναφορικά με την διαχείριση των εν λόγω δικτύων, αλλά εισαγάγουν και κάποιες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες χρήνουν όπως θα έπρεπε να ισχύουν πέραν ε, των ορίων των δικτύων τα οποία ρυθμίζονται μέσω των ε, οδηγιών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το στις ε, τοπικές αρχές, διότι αυτοί είναι κανόνες ε, που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να δεσμευτούν στο να τηρούν. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια οδηγία να την ψηφίζουμε και να συμμετέχουμε στην κατάρτιση οδηγίας για τα ευρωπαϊκά δικτύα και έπειτα να συμπεριφερόμαστε με τρόπο εντελώς αντίθετο από αυτόν που επιβάλλουν οι ε, λόγω Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι καθήκον μας να το πράξουμε και θα το πράξουμε. Όσοι εξέφρασαν την... Και η Κομισιόν εξέφρασε την λύπη της για το ότι δεν μπορεί να δώσει πιο απτές ε, ε, εξηγήσεις και να κάνει πιο απτές προτάσεις. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη αναφορά, την υπαριθμόν 27 στην ίδια διάταξη του κυρίου Θεόδωρου Δαλμάρη. Ο αναφέρον ε, δεν ε, παρευρίσκεται μεταξύ μας. Δώσω το λόγο στην πρόσφατη Κομισιόν Γκούντρουν Γκάλοφ. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά την υγεία των τροφίμων. Ο αναφέρον καταγγείλει συγκεκριμένη περίπτωση μη σεβασμού τους ε, σάδες τροφίμων στην Ελλάδα. Υποθέτω ότι σε γενικέ γραμμέ γνωρίζει η Επιτροπή σα το ιστορικό αυτή τη αναφορά. Θα ήθελα να ε, σα αναφέρω περιληπτικά. Εκτό από την αναφορά αυτή, πήρε η Κομισιόν και μία ίδια θα έλεγα ε, καταγγελία που επιβεβαιώνει τα στοιχεία που υπάρχουν στην αναφορά. Κοντά στην Αθήνα βρίσκεται μια μεγάλη αγορά που είναι και κρεατογορά, από ό,τι κατάλαβα και στην αγορά αυτή δεν τηρούνται οι κοινοτικοί κανόνες υγιεινής τροφίμων. Αυτές, ε, το αυτό παρακολουθείται από το 2006 ήδη. Έχουμε τον κανονισμό 854 που προβλέπει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τους απαραίτητους ενέχους και δεύτερον ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να κλείνουν ή να εγκρίνουν ανάλογα τι, ένα κατάστημα ή ένα σημείο πώληση βάσει των διατάξεων της, ε, του λόγου κανονισμού. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ε, θα πρέπει να αναλυφθούν περαιτέρω μέτρα. Ως Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθούμε την κατάσταση από το 2006 με μια σειρά επιθεωρήσεων όπου πραγματικά είδαμε ότι δεν τηρείται ο λόγω κανονισμός. Κατόπιν καλέσαμε την ελληνική κυβέρνηση βάσει της συνήθου διαδικασίας να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση στην κρεταγορά αυτή. Μας δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις, εγγυήσεις. Μας είπαν ότι θα υπάρχουν νέα κτίρια που θα πληρούν καλύτερα τις προϋποθέσεις. Στείλαμε και διάφορες επιστολές στην ε, ελληνική κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες, όχι μόνο σε σχέση με τις επιθεωρήσεις, αλλά και επίσημες επιστολές. Ε, πάντα ακούγαμε διάφορες εγγυήσεις, υποχωρήσεις. Η ε, τελευταία λύση και η κυρία Βασιλείου, η Επίτροπος κατά μία επίσκεψη στην Ελλάδα, τόνισε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Έγινε μετά παρατέρω επιθεώρηση για να δούμε κατά πόσον έχει διορθωθεί η κατάσταση ή όχι, σύμφωνα με τις υποσχέσεις, και είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις, Κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές φαίνεται μετακόμισαν σε ένα νέο κτίριο, αλλά καταρχήν έχουμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιμένει ούτε το ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε κρέα στην αγορά αυτή να τηρούν απαραίτητο ε, τους ε, υγειονομικούς κανόνες της Ένωσης, ούτε επιβάλλει τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τη χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας και επίσης εάν υπάρχουν καταπατήσεις ε, του, της οδηγίας αυτής, δεν υιοθετούν συγκεκριμένα μέτρα. Με δύο λόγια, η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 226 της συνθήκης. για να βρεθεί μια λύση για την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε με τη διαδικασία επιπαραβάση που ξεκινάει με την επιστολή κοινοποίηση όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει. και ίσως να καταδείξει ότι ακολουθεί με κάποια διαφορετική όδος ίσως μια που άλλαξε η κυβέρνηση στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Εάν όχι, δεν βλέπουμε καμιά άλλη δυνατότητα παρά να προχωρήσουμε με τη διαδικασία επί παραβάση. Ο κύριος Μελάς. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις ελληνικές θέσεις όσοι έχουν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε πάρει από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ειδικότερα τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, ο οποίος ήταν και ο ε, υπεύθυνος και αρμόδιος για του συγκεκριμένου προγράμματος αναβάθμισης της αγοράς, η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής. Η χονδρική διακίνηση του κρέατος σχεδόν στο σύνολό της γίνεται πλέον στις εγκαταστάσεις της νέας αγοράς και ειδικότερα στα δύο νέα συγκροτήματα κτηρίων όπου δραστηριοποιούνται 25 από τις 32 παλαιότερα εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος η έγκριση των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 8, το 2008. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η επάρκεια υποδομών και σχεδιασμού των εγκαταστάσεων της νέας αγοράς καθώς και η παράλληλη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου βασισμένου στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου με κρίσιμα σημεία ελέγχου, HASP, καλύπτουν απόλυτα τα σύγχρονα υγειονομικά και λειτουργικά πρότυπα των απαιτήσεων της κοινοτική νομοθεσίας, κάτι που θα μπορεί να γίνει και σαφές και εμφανές απόλυτα σε μια ε, επερχόμενη αποστολή των ε, υπηρεσιών της Επιτροπής στην αγορά του Ρέντι. Στην παλιά αγορά αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει μόνο 7 επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουν μετακινηθεί στα νέα κτίρια σε συνέχεια εσωτερικών ανακατατάξεων και αποχωρήσεων κάποιων επιχειρήσεων που λόγω κρίσης ούτως ή άλλως κλείσαν και φεύγουν, αποχωρούν ως νομικές μορφές από την αγορά, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια έχουν ήδη κατεδαφιστεί διευκρινίζεται για μια ακόμη φορά ότι η διάρθρωση και η υποδομή των υφιστάμενων καταστημάτων, των λίγων υφιστάμενων καταστημάτων των 7 στην παλιά αγορά του Ρέντι, που είχε προκύψει ως αποτέλεσμα εφαρμογής προγράμματος επίγουσας αναβάθμισης των καταστημάτων αυτών, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο ανάγκες χονδρικής εμπορίας κρέατος και όχι τεμαχισμού. Και το τονίζω το συγκεκριμένο γιατί θα πρέπει να ληφθεί η παράμετρος ως έχει και οποιασδήποτε ελλείψεις, τυχόν ελλείψεις, να συναρτώνται λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι τον τεμαχισμό που έχει επιπρόσθετες υγειονομικές απαιτήσει. Επισημαίνεται επίσης ότι ο χώρος της παλαιάς αγοράς μέχρι την ολοκλήρωση της νέας και αναφέρομαι στο παρελθόν και όχι στη δεδομένη χρονική στιγμή τώρα αποτελούσε χώρο ο οποίος ήταν απόλυτα ελεγχόμενος σχετικά με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων, των συνθήκων μεταφοράς, των διαμόρφωσης τιμών, της διαμόρφωσης των τιμών, με καθημερινή παρουσία των ελεγκτικών αρχών, κατά πλήρη υπέρβαση της συχνότητας που υπαγορεύει η ανάλυση επικινδυνότητας και η κατηγοριοποίηση αυτού του είδους των επιχειρήσεων, και αυτό γιατί πρόκειται για μια δέσμευση που έπρεπε να τηρήσει η χώρα, που είχαν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας, έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής. Επιπρόσθετα, επειδή υπάρχει στη συγκεκριμένη αναφορά το Δημοτικό Σφαγείο της Πρέβεζας, πρέπει να τονιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές προέβησαν σε οριστική ανάκληση της άδειας, της άδειας λειτουργίας του εν λόγω σφαγείου από τις 22 Εβδόμου το 2002. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρούμε ότι οι ισχυρισμοί της καταγγελίας στη δεδομένη χρονική στιγμή και με τη δεδομένη δομή που υπάρχει δεν έχουν κάποιο έρισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο. Ε, έχω την εντύπωση ότι ε, ικανοποιητικές φαίνονται όσα ε, οι διατυπώσεις ε, οι πρόσφατες. Ε, βεβαίως μπορούμε να αφήσουμε την υπόθεση ανοιχτή ε, αν έχουμε και νέα στοιχεία. Είμαστε ανοιχτοί ακόμα και σε επίσκεψη φαντάζομαι. Ε, πολύ ευχαριστώ κύριε Μελάκα. Να είστε καλά. Επόμενη ανακοίνωση αναφορά της ε, κυρίας ε, Lucy Jane Marie Stewart από την Βρετανία που αφορά στην, ε, στο δικαίωμά της να παίρνει σύνταξη αναπηρίας επειδή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό το οποίο είναι υπήκος. Η κυρία Στιούαρτ είναι παρούσα. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι λούση Στιούαρτ, είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και Ευρωπαίος πολίτης. Μπορώ να έχω παρακαλώ τα λεφτά μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινή Στιούαρτ. Ε, από τη μεριά της Επιτροπής. Είμαι η μητέρα της Λούση και είμαι πολύ περήφανη που η όμορφη αυτή είναι κοπέλα είναι η κόρη μου. Το μόνο το οποίο ζητάει είναι αυτό που ζητάει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης. Μια ζωή, ένα σπίτι, μια δουλειά, καμία διάκριση και θα πρέπει να μπορεί να υποφελείται των δικαιωμάτων της όχι μόνο στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά και στα πλαίσια της βρετανικής νομοθεσίας. Έχω στείλει τα απαραίτητα έγγραφα, η Επιτροπή σας και οι μεμονωμένοι βουλευτές έχουν λάβει τα έγγραφα αυτά. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Θα ήθελα να σας διαβάσω μία επιστολή που αποστάλει προς την ε, κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου για την ε, περίπτωση της Λούση. Το 2002 ο τότε Υπουργός Τζακ Στρό είχε πει στην ε, Επιτροπή ότι ε, θα μπορούσε η ε, Τζέιν να λάβει τα επιδόματα αυτά, ότι θα μπορούσαν τελικά να τις επιστρέψουν, αν θέλετε, αναδρομικά και τα χρήματα τα οποία της όφυλαν, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε στη συνέχεια. Η επιστολή αυτή είναι του Φεβρουαρίου του 2009 και λέγεται από τον Ευρωβουλευτή προς την κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου ότι η Λούση Στούαρτ παίρνει επίδομα αναπηρίας κανονικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο της δίδεται από τον έκτο μήνα της ζωής της. Σύμφωνα με την νομοθεσία 1247-92 με την νομοθεσία του 1971 επίσης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επίδομα αναπηρίας και κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην ε, Ισπανία. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την ε, προσοχή σας στην περίπτωση παράβασης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2002, ιδίω των διατάξεων που εφαρμόζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και αναφέρεται επίσης στην ανταλλαγή επιστολών που έγινε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου καθίσταται σαφές ότι η Lucy Τζέιν θα πρέπει βάσει της κοινοτική νομοθεσία να λαμβάνει τα επιδόματα αναπηρία τα οποία τη ε, δινόντουσαν στον Ηνωμένο Βασίλειο προτού μετακομίσει στην Ισπανία. Επίση, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνειδητοποιεί ποιε είναι οι επιπτώσει από την εφαρμογή αποφάσεων του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ανάλογες υποθέσεις που έχουν εξεταστεί από το δικαστήριο αυτό και όπου έχει ζητηθεί κάθε φορά η ίση μεταχείριση καθώς επίσης και η εφαρμογή του κανονισμού 1408 του 71. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεχή υποβολή του επιδόματος αναπηρίας και μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε ότι και ο οποιοδήποτε άλλος ετών στο μέλλον, στην ίδια περίπτωση δηλαδή όπως και η Λούση, θα χαίρει των ίδιων δικαιωμάτων. Βάσει λοιπόν των δεσμεύσεων αυτών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε την περίπτωση παραβίασης στην, στην υπόθεση C. Παύλα 2002-49. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε ανώτερο δικαστήριο. Έχετε ήδη το σχέδιο απόφασης το οποίο θα πάει στο ΔΕΚ. Η νέα όμως νομοθεσία οι νέες ρυθμίσεις που ισχύουν στην Αγγλία προβλέπουν ότι μπορούν κάποιες ε, δικαστικές υποθέσεις να συνδυαστούν με άλλες ανάλογες υποθέσεις και να παρουσιαστούν από κοινού. Η περίπτωση της ε, Λούση όμως έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Ε, την Επιτροπή σας έχει υποβληθεί και στα πλαίσια άλλης αναφοράς στο παρελθόν. Έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με τους ε, ευρωβουλευτές της δικής μου περιφέρειας, δεν έλαβα όμως μια απάντηση. Προσπάθησα να ασκήσω πίεση, κάποιοι μου είπαν ότι θα πρέπει να πάρω τα χρήματα από την Ισπανία. Κάποιος άλλος μου είπε ότι ε, δεν ανήκεται στους εκλογείς μου. Ο κύριος Βάτσον ε, μόνο τελικά με βοήθησε, ο οποίος δεν είναι και άμεσα, θέλετε, δικός μου ευρωβουλευτής αυτό είναι απόλυτη ντροπή που είναι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ, που είναι οι ευρωβουλευτέ τη εκλογική μου περιφέρεια. Αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να δώσω μόνο μια μάχη για την κόρη μου και εκπροσωπώντα και του υπόλοιπου ανάπηρου στον Ηνωμένο Βασίλειο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Εγώ σα ευχαριστώ, κυρία. Θα περιμέ... Πρώτα να μιλήσει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή και μετά εσεί, κύριε Βότσον. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Στιούαρτ ε, που εξήγησε την υπόθεση της κόρης της Λούση και την Λούση για την παρέμβασή της. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε δύο περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε την διαμαρτυρία της κυρίας Στιούαρτ αναφορικά με την άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να καταβάλει στην Λούση το επίδομα αναπηρίας και θεωρούμε πως αυτή η άρνηση είναι αντίθετη με το άρθρο 3 του κανονισμού 1408-71 το οποίο αφορά στην ίση μεταχείριση και η άρνηση του Βασιλείου να εξαγάγει αυτό το επίδομα είναι επίσης αντίθετο από την αρχή της μεταχείρισης ε, ήρθαμε σε επαφή με τις ε, αρχές του Ινωμένου Βασιλείου και μας απάντησαν ότι δεν είναι σε θέση να μας δώσουν περαιτέρω προφορίες διότι η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Μετά από αυτή την απάντηση ξεκινήσαμε διαδικασία επί παραβάση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ω εκ τούτου προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω περαιτέρω προφορίες περί αυτού. Αλλά περιπτώσει παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ ε, την υπόθεση και δεν χάνουμε χρόνο. Και το δεύτερο σημείο που ανέφερε η κυρία Στιούαρπ για την διαδικασία παραβίασης το 2002 ε, ολοκληρώθηκε το 2004. Κλείσαμε την υπόθεση αυτή διότι η επίσημη απάντηση των αρχών του Νομού Βασιλείου ανέφερε ότι αυτό το επίδομα δεν χορηγείται στους ε, υπηκόους που κατοικούν στο εξωτερικό. Αποφασίσαμε να κλείσουμε την υπόθεση στην περίπτωση αυτή, αλλά φυσικά αν υπάρχουν ε, προβλήματα θα το επανεξετάσουμε το ζήτημα. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις και για τη δράση και τους ε, ζητάω να συνεχίσουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται η υπόθεση αυτή στην Επιτροπή. Θα έφτασε το 2002. Η κυβέρνηση των Βασιλείου υποσχέθηκε να τροποποιήσει τον ε, νόμο, αλλά δεν το έπραξε και έτσι η Λούστη δεν μπορεί να λάβει την ανταποδοτική παροχή αναπηρίας. Ισχυρίζεται ότι δεν δικαιούται τον Βασίλειο αυτής της ε, παροχή, διότι δεν κατοικεί στον Βασίλειο πριν από την υποβολή και μετά αλλά η κυρία Στιούαρτ ε, είπε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 1408 71 δικαιούται αυτού του επιδόματο. Η περίπτωση αυτή βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον λόγο λοιπόν αυτό η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θέλει να δώσει περαιτέρω προφορίε να πάρει μια επίσημη θέση. Πάντω η Κομισιόν έχει απόλυτο δίκιο που επικέντρωσε το, στο άρθρο 3 του κανονισμού 1408 71 διότι δηλαδή δικαιούται η Λούση Στιούαρτ παρόμοιο επίδομα. Η κυρία Στιούαρτ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ε, προσέγγισε έναν βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας και εκπλήσωμε που ο κύριος Χάναν ε, απάντησε ότι δεν μπορεί να τη βοηθήσει και ανήκει στη συντηρητική ομάδα. Ε, θεωρεί ότι κάποιος δεν θα πρέπει να ζητάει παροχές αφού έχει καταλήψει την χώρα. Νομίζω ότι καθήκον του κ. Χάναν είναι να ε, βοηθήσει την κυρία Στιούαρτ, ε, της οποίας η κόρη έχει πέσει θύμα μιας εσφαλμένης ερμηνείας ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν με τα χαράς να βοηθήσω την κυρία Στιούαρτ θεωρώ πως η κόρη της είναι, έχει πέσει θύμα αδικίας, κατάφορης και ελπίζουμε η κατάσταση να επανορθωθεί και ζητώ από την Κομισιόν να συνεχίσει τις προσπάθειές της εξονόμερος της Λούση Στιούαρτ. Κύριε Βότσον, είναι πραγματικά εντυπωσιακό <laughs> πώς μπορεί να είναι τόσο εμφανές και να μην ε, είναι νόμιμη η στάση του κράτους απέναντι στις υποχρεώσεις ενός Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί η Λούση είναι Ευρωπαία πολίτης, δεν είναι μόνον πολίτης της Μεγάλης Βρετανίας εμείς μπορούμε να γράψουμε ε, μια επιστολή, να συντάξουμε μια επιστολή στον Υπουργό, τον Άγγλο, για το θέμα, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο υπέρ του αιτήματο της ε, Λούση και της μητέρα της. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το επόμενο που αφορά, μισό λεπτό, αφορά την ε, ε, την αναφορά του κυρίου Άγγελ Λάσεφ από την Βουλγαρία ε, για τη Συντονιστική Επιτροπή ε, για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην πόλη Νόβη Ισκάρ με 1920 υπογραφές σχετικά με την καταστροφική ρήπανση του προαστίου Νόβη Ισκάρ της Σόφιας λόγω επικίνδυνων αποβλήτων. Από τη μεριά του, της Επιτροπής η κυρία Λουτμίλα Πόποβα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας απαντήσω στα αγγλικά για την ε, αναφορά αυτή. Πράγματι, ε, πήραμε πληροφορίες ε, όσον αφορά αυτό το θέμα της αναφοράς το 2008. Οι πληροφορίες που πήραμε ήταν εντυπωσιακέ. και αμέσω ήρθε την προσοχή μας και ήρθαμε σε επαφή με τι βουλευτικέ αρχές για να πάρουμε πληροφορίε. Φαίνεται ότι πράγματι κάποια εταιρεία είχε παράνομα εγκαταστήσει εκεί κάποια απόβλητα οικοδομών, παρόλο που δεν πρόκειται για χωματερή, η αντίδραση της Κομισιόν οδήγησε σε αντίδραση της εθνικής κυβέρνησης τελικά αυτή τη στιγμή το ίμιση των αποβλήτων αυτών των μπαζών έχει αποσυρθεί και συνεχίζεται η απόσυρση γιατί η ποσότητα που είχε αποτεθεί εκεί είναι τεράστια. Ακόμα δεν έχουν ε, έρθει σε επαφή μαζί μας οι ε, αναφέροντες. Άρα έχουμε την εντύπωση ότι μάλλον ικανοποιήθηκαν από την κατάσταση και ότι περιμένουν να ολοκληρωθεί η απόσταση αυτή. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και μηνύα ζητάμε πληροφορίες από τις Εθνικές Αρχές της Βουλγαρίας όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται. τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή την τελευταία φορά που πήραμε τις ε, πληροφορίες και σύμφωνα με τα τελευταίες πληροφορίες περίπου 400.000 τόνοι ε, αποβλήτων έχουν αποσυρθεί. Η κατάσταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχει επιληθεί πλήρως, αλλά παραμένουμε στην παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Ίσως είναι από τις αισιόδοξε στιγμέ αυτής της συνεδρίας ότι έχουμε αποτελεσματικότητα στις δράσεις μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πόποβα. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Περιμένουμε... All close the case. or follow up? All ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναπροκύψει το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ε, αναφορά της κυρίας Εύα Σίνκεβιτς από την Πολωνία για την περιβαλλοντολογική οργάνωση σχετικά με τη ρήπανση που οφείλεται σε απόβλητα από την επεξεργασία νεκρών ζώων. Από τη μεριά της ε, Επιτροπής, ο κύριος Κούστερ. Ο κύριος Κούστερ, παρακαλώ. Thank you, Madam Chairman. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Η παρουσίασή μας έχει δύο στοιχεία. Η μία την προστασία της δημόσιας και η άλλη προστασία του περιβάλλοντος από τη μόνηση. Η αναφορά που μας ε, μετεβάστη ε, συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία όσον αφορά την ε, ταφή ζώων Πρόκειται που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, που έχουν ψοφήσει φερρυπίν. Η αναφορά περιλαμβάνει διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά τις επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό γύρω από την κατάσταση αυτή που δυστυχώς δεν επίπτυξε στην οδηγία 100, 1772 ε, δύο που αφορά ακριβώ τη δυνατότητα της αποφυγής της ε, μεταβίβασης ε, επιζωτιών και ασθενειών στους κατοίκους. Δηλαδή το αντικείμενο της οδηγίας αυτής είναι να αντιμετωπιστούν τα ε, υποπροϊόντα αυτών των ζώων κατά τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες ε, πτυχές όσον αφορά την μονάδα αυτή επεξεργασία στην Πολωνία. Η μία πτυχή λέει ότι είναι παράνομο το εργοστάσιο. Αλλά σύμφωνα με τη δική μας ε, έρευνα έχουν ληφθεί απαραίτητε απαραίτητες άδειες ε, για την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων. Άλλες ε, προσφυγές αφορούν την χρήση του τελικού προϊόντος της εταιρείας αυτής, δηλαδή ως αλεύρων και κρεαταλεύρων, γιατί παραδείγματος χάρη τα νεκρά αυτά ζώα δεν μεταφέρονται κατεψυγμένα. Μία τέτοια μονάδα εργασίας πρέπει να είναι συμμορφωμένη με κάποιες βασικές αρχές ε, για την προστασία της υγείας και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ασφαλές. Όσον αφορά τα οργανικά λιπάσματα, η οδηγία απαγορεύει να χρησιμοποιείται σε, ε, ζω, σε τόπους ε, βοσκής, αλλά επιτρέπει να χρησιμοποιείται αλλού όταν ληφθούν οι απαραίτητες ε, προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις επιτόπου όσον αφορά την ταφή των νεκρών ζώων, η οδηγία δεν προβλέπει την ε, ταφή των νεκρών ζώων. Στο παρελθόν υπήρχε κάτι τέτοιο στην οδηγία αυτή, αλλά όχι πια. Από το 2002 δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Και επίσης η ταφή των νεκρών Ζών επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών. Παραδείγματος χάρη σε περίπτωση επιζωοτία. Και είναι καλύτερο στην περίπτωση να ταφούν επιτόπου παρά να μεταφερθούν. Όσον αφορά τώρα την μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, η οδηγία είναι σαφής. Λέει ότι θα πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά οχήματα. Από την άλλη μεριά δεν διευκρινίζει η οδηγία ότι θα πρέπει να είναι κατεψυγμένα τα υποπροϊόντα αυτά. Εκτός αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πολύ συγκεκριμένες ε, χρήσεις, παραδείγματο χάρη για την παραγωγή ζωοτροφών. Εμείς θα προωθήσουμε τις πληροφορίες στην υπηρεσία κτηνοτροφικών ελέγχων που βρίσκεται στην Ιρλανδία και που κάνει τακτικές έρευνες στα κράτη-μέλη. Γιατί κάποια από τα στοιχεία της ε, αναφοράς ίσως είναι καλό να ελεγχθούν την επόμενη φορά που η υπηρεσία αυτή θα πάει στην Πολωνία. Όσον αφορά τώρα το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτό, αλλά από ό,τι είδα στην απάντηση τη γενική διεύθυνση Περιβάλλοντος, λείπουν από την αναφορά κάποια στοιχεία για να μπορέσει πραγματικά να ε, εξεταστεί κατά πόσο πρόκειται για παραβίαση του κοινωνικής νομοθεσία ή όχι. Και κατά πόσο να απειλούνται προστατευόμενε περιοχές. Ευχαριστώ. Πολύ. Κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να παρέμβει. Ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια <clears throat> ασάφεια στις διατυπώσεις της Επιτροπής. Ε, δεν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τις κατηγορίες για τις δυσμενείς συνέπειες των θαμένων ζώων στα υπόγεια ύδατα. Δεν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε παραβίαση της οδηγίας ε, δεν το καταλαβαίνω ομολογώ. Ποιος μπορεί να είναι σε θέση να το κάνει. There Υπάρχουν πολλά στοιχεία σε αυτή την αναφορά, Πρόεδρε. Καμιά φορά τα σημεία αυτά αφορούν τη συμμόρφωση ημί με την κοινοτική νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη, κατά πόσον η βιομηχανική αυτή εγκατάσταση έχει άδεια ή δεν έχει άδεια για να ασκήσει τι δραστηριότητε που ασχεί. Άλλα θέματα αναφέρονται στο γεγονός ότι τα οχήματα αυτά στάζουν. Αυτό είναι ίσως μια γενική ε, αναφορά, ε, αλλά δεν αναφέρονται στη συμμόρφωση ή μη με κάποια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Γι' αυτό είχαμε την εντύπωση ότι θα ήταν καλό να μελετηθεί το θέμα επιτόπου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους διάφορους παράγοντες και να γίνει κάποια επιθεώρηση επιτόπου η, η οποία είναι κάλλιστα δυνατόν να γίνει. Ούτω ώστε οι επιθεωρητέ που θα πάνε εκεί θα λάβουν υπόψη και τον κοινοτικό και αλλά και το τι συμβαίνει επί τόπου, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και έτσι θα μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να γίνει καλύτερη αξιολόγηση του θέματο. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ελπίζω ότι θα συγκροτηθεί σύντομα η Επιτροπή, ότι θα έχουμε τα αποτελέσματά της. Επομένως κρατούμε την αναφορά ανοιχτή, την περίπτωση ανοιχτή, για να την ξανασυζητήσουμε όταν έχουμε περισσότερα δεδομένα από τη μεριά της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στην τράπεζα, και την παραβίαση της Οδηγίας 2002-14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Συμβουλίου της Ευρώπης το 2002 ε, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωση και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο κύριος Δημητρίου από την μεριά της Επιτροπής. Ναι. Ευχαριστώ. Ε, thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ανακοίνωση των υπηρεσιών της Κομισιόν σχετικά με την αναφορά αυτή υπευλήθη το 2008 στην Επιτροπή σας και αναφέρει λεπτομεριακά τα γεγονότα και την πρώτη προσέγγιση της Κομισιόν σχετικά με την αναφορά αυτή. Μετά από αυτή την πρώτη ανακοίνωση, οι υπηρεσίε της Κομισιόν συνέταξαν μια συρωματική ανακοίνωση το Μάρτιο 2009, αλλά για κάποιους ε, μυστήριους ε, λόγους ε, δεν έφτασε πότε στην Επιτροπή σας η ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Κομισιόν συνέταξαν μια νέα ενημερωμένη ανακοίνωση στις αρχές Οκτωβρίου, πριν από ένα μήνα, που ελπίζουμε να σας διαβαστεί συντόμως. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω σχετικά με τις εξελίξεις. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι πως ο αναφέρον έχει υποβάλει και προς την Κομισιόν μια επίσημη διαμαρτυρία που αφορά στα ίδια γεγονότα. Αυτό λοιπόν το έχει, έχει καταγραφεί από τη Γενική Γραμματεία της Κομισιόν και εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή η αναφορά, όπως και η διαμαρτυρία, αναφέρεται σε δύο χωριστά ζητήματα. Το ένα αφορά την οδηγία 2002-14, την οδηγία που αφορά την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή κοινότητα και το δεύτερο που αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού και δι των κρατικών ενισχύσεων. Θα ήθελα να σας δώσω πληροφορίες τώρα σχετικά με το πρώτο θέμα, δηλαδή την ε, παραβίαση της 2002-2014 και μετά δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που θα σας ενημερώσει για το θέμα ε, που άπτεται της πτυχής του ανταγωνισμού. μια που έχει καταχωρηθεί και ως ε, επίσημη διαμαρτυρία, της Κομισιόν ε, ήρθαν ε, επανειλημμένα σε επαφές πρώτα απ' όλα με τις ελληνικές αρχές και δεύτερον με τον αναφέροντα και ειδικά τον νομικό του εκπρόσωπο. Στην πρώτη ανακοίνωση της Κομισιόν το 2008 σας ενημερώνουμε πως η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές τον Ιανουάριο 2008 μέσω επιστολής όπου μας απάντησαν τον Μάρτιο 2008 οι ελληνικές αρχές. Μετά αυτήν την ανταλλαγή επιστολών, οι υπηρεσίε του Κομισιόν ήρθαν σε επαφή με τον αναφέροντα και τον υποβάλλοντα τη διαμαρτυρία. Ε, έλαβε κάποιες ε, απαντήσεις ε, και η Κομισιόν κατέληξε μετά από ενδελεχή έλεγχο των γεγονότων και των στοιχείων ότι όντως υπήρχε πρόβλημα όχι σε ό,τι αφορά την μεταφορά της οδηγίας 2002-2014 στην Ελλάδα, αλλά σχετικά με την εφαρμογή της στην πράξη και στο συγκεκριμένο κλάδο. Η οδηγία 2002-14 μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με προεδρικό διάταγμα 2.14 του 2006. 2040, συγγνώμη, του 2006. Και σε αυτό το προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ένα μεγάλο κομμάτι των διατάξεων της οδηγίας. Αυτό το οποίο δικαιωόταν εδώ ήταν η ερμηνεία από πλευρά ελληνικών αρχών αυτή τη ε, οδηγία. Οι ελληνικέ αρχέ ε, ισχυρίστηκαν σε πρώτη φάση ότι η οδηγία 2012-2014 δεν ε, εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και ως επιχείρημα ανέφεραν πως το θέμα αυτό αφορά θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δεν καλύπτεται από τις ε, πρόνοιες της οδηγίας. Οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι της αυτής άποψης και έτσι τη 17 Οκτωβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαβίβασε στις ελληνικές αρχές μια επιστολή η οποία αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα ε, σε ό,τι φορά την εφαρμογή του κοινωτικού, της κοινωνικής νομοθεσίας, ειδικά σε ό,τι φορά την οδηγία 2014 και κάλεσε ως ήθιστε τις ελληνικές αρχές ε, να λάβουν θέση. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 16 Δεκεμβρίου 2008 επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα που είχαν αναφέρει στην προηγούμενη επιστολή τους ε, λέγοντας ε, πως ε, η υπόθεση αυτή δεν καλύπτεται από την οδηγία 2002-14. Αλλά η Κομισιόν δεν επίθη και εξέδωσε γνώμη που έβαλε στις 26 Ιουνίου 2009 προς τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αιτιολογημένη γνώμη, οι Ελληνικέ αρχές απάντησαν ε, με επιστολή 12 ε, Αυγούστου 2009. Σε αυτή την επιστολή οι ελληνικέ αρχές συμφώνησαν με την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφώνησαν ότι η Οδηγία 2002-114 ε, έπρεπε να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση και η υπάλληλοι των ε, τραπεζών θα έπρεπε να ενημερώνονται από τον εργοδότη του σχετικά με τι προθέσεις ε, να υποβάλουν ε, στο ΕΤΑΤ το αίτημα για τη συντήρηση των εργαζομένων σε αυτό το ταμείο, το νέο Ταμείο Ασφάλιση των Τραπεζοπαλλήλων. Αυτό που έχει σημασία είναι πως οι ελληνικές αρχές ε, στην επιστολή 12 Αυγούστου 2009 ε, είχαν προσαρτήσει και μια εγκύκλιο προς το οποίο αφορά στο Υπουργείο Κοινωνική Προστασία. Αυτή η εγκύκλιο ανακοινώθηκε προ όλε τι αρμόδιε ελληνικέ αρχέ, ιδιαίτερα στην επιθεώρηση εργασία και αλλά επίσης και σε άλλους ενδιαφερομένους όπως συνδικαλιστικέ οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Αυτή η εγκύκλειος αναφέρει τις υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με θέματα ενημέρωσης και διαβούλευση των εργαζομένων, όπως επίσης και την εφαρμογή του, μάλλον και την δυνατότητα της εργασίας να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης ε, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις ε, περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων. Περαιτέρω, ως ήθιστε, οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσαν ε, τον ενάγοντα και τον αναφέροντα με επιστολή της 9ης Σεπτεμβρίου 2009. Σε αυτή την επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τον Νάγοντα για τη νέα ε, θέση των ελληνικών αρχών περί του θέματος και προστάτησε επίσης και την ε, ερμηνευτική εγκύκλιο. Ως ήθιστε και εδώ, η Κομισιόν ζήτησε από τον Ενάγοντα να υποβάλει ενδεχόμενα σχόλιά του και τον ενημέρωσε επίσης σχετικά με την πρόθεσή της ε, να κλείσει την υπόθεση σε περίπτωση που δεν υποβάλλει περαιτέρω προφορίες ε, ή και σχόλια. Ο Ενάγων δεν υπέβαλε κανένα σχόλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και το κλείσιμο της υπόθεσης ε, μερικές μέρες αργότερα, δηλαδή συγκεκριμένα την 29η Οκτωβρίου 2009. Δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφό μου ειδικά με την πτυχή της, ε, του ανταγωνισμού και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Όσον αφορά το άλλο τμήμα της αναφοράς, δηλαδή την ε, κρατική ενίσχυση στην περίπτωση της Αλφα θα ήθελα να σας υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε πει και στην πρώτη μας επιστολή που στείλαμε προς την Επιτροπή Αναφορών. το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πάρει μια απόφαση όσον αφορά την μεταφορά συνταξι... Ε, δικαιωμάτων συντάξεων στα πλαίσια του τραπεζικού τομέα. Είχαμε πει ότι ακολουθεί το τότε η ελληνική εθνική νομοθεσία που ίσχυε προφανώς και για την Αλφα Bank. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα είχε πει ότι η μεταφορά των επιπλέον συνταξιδοτικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. επομένως δεν τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού ακόμα ε, εφόσον ακολουθηθούν ε, βέβαια οι διατάξεις της α, ε, σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση τώρα της Αλφα Bank, η μεταφορά των, νέων, των επιπλέον αυτών δικαιωμάτων βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Η, Ευρωπαϊκή, η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επομένω εξακολουθεί και ισχύει. Ο Σύλλογο των Εργαζομένων τη ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ μα λέει βέβαια τώρα ότι πιστεύουν ότι τίθεται ζήτημα κρατική ενίσχυση και ότι η ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ θα πρέπει να καταβάλει λιγότερα από ότι καταβάλει μάλλον λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε να καταβάλει. Έχουμε όμω απαραίτητε πληροφορίε στα χέρια μα και δεν μα έχουν δοθεί νέα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν έχει γίνει σεβαστή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 ενημερώσαμε καταλήλως τον αναφέροντα που είναι και προσφεύγων και του ζητήσαμε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες που να καταδεικνύουν τελικά με ποιο τρόπο η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έγινε σεβαστή, δεν τηρήθηκε από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές. Δεν μας δόθηκε όμως η απάντηση αυτή, δεν μας δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες που ζητήσαμε. Αξιολογήσαμε λοιπόν την κατάσταση και εφόσον ισχύει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούμε ότι αν ο ενάγων δεν μας δώσει απτά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει γίνει σεβαστή απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις εθνικές νομοθεσίες, τότε η καταγγελία αυτή δεν έχει λόγο να μείνει πλέον ανοιχτή, μπορεί να κλείσει. Έχει ακόμα δύο-τρει εβδομάδε ο ενάγων προκειμένου να δώσει περισσότερα στοιχεία. Αν δεν λάβουμε τα στοιχεία αυτά, θα κλείσει το ζήτημα. Όσον αφορά το τμήμα της κρατικής ενίσχυσης, τη καζόμενη κρατική ενίσχυση. Ευχαριστώ. Ε, ε, περιμένουμε νεότερα, αν χρειαστεί να κλείσει όχι. Ευχαριστούμε ε, πολύ. Ε, του κυρίου είναι η παρικμόν 32 του κυρίου Φραγκάκη ε, για το δικηγορικό γραφείο Σουριαδάκης, Φραγκάκης, Καλτσάς και Παντελάκης σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ε, είναι εδώ, ελπίζω, από την Επιτροπή η κυρία Εύα Thank you, ε, thank you, Mrs. Chairman. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα βασικά επιχειρήματα που έχουμε στην αναφορά αυτή έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδας σε ένα ενιαίο Ταμείο Ασφάλειας, Ασφάλισης Μισθωτών και εικάζονται εδώ πέρα ότι έχουν γίνει διάφορες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας μέσω δηλαδή της ελληνικής νομοθεσίας που εγκρίθηκε. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα στην αφορά αυτή αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας, η οποία έκλεισε πρόσφατα και έχουν εξηγηθεί οι περιπτώσεις αυτές, οι περιστάσεις αυτές σε μια ανταλλαγή επιστολών που είχαμε με τον Ενάγοντα, όπου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση. Τα βασικά επιχειρήματα, τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στην αναφορά εξετάστηκαν σε σχέση με την ε, απαγόρευση της νομισματικής ε, χρηματοδότησης σε σχέση με την ε, ανεξαρτησία της Τράπεζας Ελλάδος και είχαν να κάνουν επίσης και με τη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, δηλαδή την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης, βάσει της αξιολόγησης που έγινε και μετά από λογιστικό έλεγχο που έγινε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε συμπέρασμα ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας, οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας δεν παραβιάζουν την υφιστάμενη απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. και επίσης δεν εντοπίστηκε παραβίαση όσον αφορά τον κανονισμό του Συμβουλίου για την ερμηνεία του άρθρου 100. του άρθρου 4 της συνθήκης. 104, με συγχωρείτε. 104β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, δηλαδή με τη διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεωρεί ότι δεν έχει υπάρξει εδώ πέρα καμία, κανένα ζήτημα παραβίασης της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως λέγεται στο άρθρο 108 της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κεντρική Τράπεζα της ότι μάλλον δεν ήρθαν σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτού γίνει η συμπερίληψη του Συλλόγου Υπαλλήλων τη Τράπεζα Ελλάδο στο Ταμείο ή ΚΑΕΤΑΜ, δεν αποτελεί παραβίαση τη κοινοτική νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζεται ότι η προσέγγιση που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση και την οποία καταγγέλει τελικά ο αναφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν συνάδει απόλυτα με το καταστατικό της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Θα έπρεπε όντως να είχε γίνει μια κάποια διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα προτού εγκριθεί η νομοθεσία αυτή. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίστηκε και στο ζήτημα της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εδώ προβλέπεται υποχρέωση διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκ των προτέρων όταν το κράτος εγκρίνει σχετική νομοθεσία. Ενώ εδώ πέρα δημοσιεύτηκε μια γνωμοδότηση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία λήφθηκε υπόψη από τις ε, ελληνικές αρχές μόνο εκ των υστέρων, αφού είχε εγκριθεί δηλαδή η εθνική νομοθεσία. Όπως είπα και πριν από λίγο, μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μία απόφαση. Προτού όμως ληφθεί η απόφαση αυτή, στείλαμε μία επιστολή στον αναφέροντα, ζητώντας του να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα έγγραφα ή κάποια παραπάνω επιχειρήματα για ποιο λόγο δηλαδή δεν θα έπρεπε να κλείσει η υπόθεση. Στην ε, επιστολή που λάβαμε τον ε, σε μια επιστολή που μας έστειλε το Μάρτιο, ο αναφέροντας επαναλήφθησαν τα αρχικά επιχειρήματα και βάσει της επιστολής αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τελικά να κλείσει την υπόθεση. Και έκλεισε τον ε, περασμένο μήνα τελικά η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ε, αν δεν υπάρχει ε, παρατήρηση. Ε, προτείνουμε το Προεδρείο να κλείσουμε με αυτήν την ε, αναφορά γιατί έχουμε υπερβεί τα όρια της παρουσίας των, <laughs> της ομάδας των διερμηνέων. Επομένως από την 33 και εξής θα πάμε στον Δεκέμβρη. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ και, τα, και τους εκπροσώπους της Επιτροπής για, τις, για την παρουσία τους εδώ. Από τον κοτσιφό, ναι, από εγώ προτείνω, ναι. επειδή είναι ο μόνο που έχει απαντήσει, γιατί στείλαμε το καλοκαίρι και τώρα απαντάει, είχε στείλει μήνυμα σε αυτόν τον Αύγουστο, εγώ είδα προχτέ τον Γουσίδη που ήταν τον παλιό ναι. πρόεδρο. Ναι, ναι. Του λέω θέλετε να την κλείσουμε ή να μην την κλείσουμε. Και φαίνεται του έβαλε. Ναι, αλλά θα αρχίσουμε αυτό το σαν Μία αναφορά. Τι άλλε θα τι κλείσουμε γιατί, δεν μα απαντάνε. Και εγώ νομίζω ότι και, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, λέει δεν υπάρχει περίπτωση γιατί η Ελλάδα έχει εφαρμόσει το, την, την νομοθεσία την στιγμή που κάποιος πολίτης έχει πρόβλημα